Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Good morning, dear guests. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, βουλευτές, ευρωβουλευτές. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασής μας και θα μιλήσω λιθουανικά. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί ομιλητές, αγαπητοί συμμετέχοντες, είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να κηρύσω την έναρξη αυτής της διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης που είναι σήμερα αφιερωμένη στην Διεθνή η ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας. Το θέμα που έχουμε επιλέξει για αυτή τη σημερινή συνεδρίαση είναι περισσότερη δύναμη στα χέρια των κοριτσιών και των γυναικών όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ε, πληροφορική. Κλειδί για το μέλλον. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν υποδεχόμαστε εδώ 27 μέλη από 17 Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας. Επίσης, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε όλους και προσβλέπουμε στις δικές σας ε, εισηγήσεις και συνεισφορές σε αυτήν την σημαντική συζήτηση. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες ανακοινώσεις για τα πρακτικά. Να ξέρετε ότι η εκδήλωση αυτή οργανώνεται σε συνεργασία με την Διεύθυνση για τις σχέσεις μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επίσης, η διερμηνία, πρέπει να ξέρετε, είναι διαθέσιμη σε όλες σχεδόν τις ε, επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τα Ιρλανδικά. Επίσης, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Στην αρχή της εκδήλωσης, δεν προβλέπεται συζήτηση γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη. Η συζήτηση θα λάβει χώρα όταν θα ακούσουμε τα πάνελ. Σημειώστε επίσης ότι ο χρόνος των παρεμβάσεων είναι περιορισμένος τόσο από τα μέλη των πάνελ όσο και από το κρατήριο. Πρέπει να τηρήσουμε την ημερήσια διάταξη προκειμένου να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε και τα θέματα. Οπότε ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη αν περιορίσω το χρόνο των ομιλητών. Τώρα, οι εθνικοί βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα από τα έτυπα τα οποία έχουν μοιράσει οι κλητήρες, οι οποίε στη συνέχεια θα τα συγκεντρώσουν και θα τα δώσουν στους συντονιστές. Το θέμα τη σημερινή μα εκδήλωση, όπω είπαμε, είναι περισσότερη δύναμη στα κορίτσια και στι γυναίκε, στα μέσα ενημέρωση και στην πληροφορική. Και ότι αυτό είναι κλειδί για το μέλλον. Πρόκειται για ένα θέμα παγκόσμιας εμβέλειας, διότι τα μέσα ενημέρωσης διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και πλαισιώνουν την πληροφορία. Συγχρόνως, οι τεχνολογίες πληροφορικής εμπλέκονται σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της κοινωνίας. Συνεπώς, τόσο τα μέσα ενημέρωσης όσο και πληροφορική έχουν τεράστιες δυνατότητες για να ενισχύσουν τις γυναίκες, να τις προωθήσουν. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση, να εκπροσωπούνται και να εμφανίζονται όπως πραγματικά είναι σε όλους αυτούς τους τομείς. Η Επιτροπή των Γυναικών λοιπόν ασχολείται όλους ιδιαίτερους με αυτά τα θέματα. Το 2016 εγκρίναμε μια έκθεση με τίτλο «Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και ενίσχυση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή». Συντάκτρια ήταν η κυρία Τέρι Ρέντκερ που θα αναλάβει και το συντονισμό του τρίτου πάνελ. Επιπλέον, πρόσφατα εγκρίναμε έκθεση για την ισότητα των δύο φύλων στο το των μέσων ενημέρωσης. Ε, συντάκτρια ήταν η κυρία Μικαέλα Σόντροβα που θα συμμετάσχει στο πρώτο πάνελ. Επίσης, ετοιμάσαμε και ένα ψήφισμα αλλά και μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ακριβώς αυτό το θέμα, την περισσότερη δύναμη δηλαδή που πρέπει να έχουν οι γυναίκες και τα κορίτσια κατά τη διάρκεια της ψηφιακής εποχής με συγγήτρια την κυρία Νιέσκα Κοσλόφσκα Ράγεβιτς που θα είναι συντονίστρια του δεύτερου πάνελ. Επίσης, να ξέρετε ότι μία αντιπροσωπεία εννέα ευρωβουλευτών υπό τη δικιά μου προεδρία θα πάμε στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχουμε εκεί στην 60 ε, δεύτερη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά το θέμα ακριβώ της θέσης της γυναίκας. Πρόκειται για τη συμμετοχή, την πρόσβαση των γυναικών στα μέσα ενημέρωση, στην πληροφορία, στις τεχνολογίες και την επίπτωση που έχει αυτή προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες να ε, αποκτήσουν περισσότερη δύναμη. Οι δικέ σας εισηγήσει και η συνεισφορά σίγουρα θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμμετέχοντες, Ελπίζαμε ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Αντώνιο Ταγιάννη, θα μπορούσε να έρθει να κηρύξει την έναρξη των εργασιών μα. Μα ενημέρωσε όμω πριν από λίγε μέρε ότι δυστυχώ δεν θα μπορέσει. Αυτό όμω που έκανε είναι ότι μα έστειλε ένα βίντεο. Βιντεογραφημένο μήνυμα δηλαδή το οποίο και θα ακούσουμε τώρα. Παρακαλώ. Καραβίλια. Αγαπητή Βίλια, αγαπητή Βέρα, αγαπητή Μαρίγια. Το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για να εξασφαλίσει σε όλες τις γυναίκες ισότητα ε, στην πραγματικότητα και δικαιώματα. Φέτος ασχολούμαστε με το θέμα της χειραφέτησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις τεχνολογίες ε, της επικοινωνίας. Το να καταφέρουμε την ισότητα του φύλου σε αυτού του ε, τομεί κλειδιά τη ε, τεχνολογική επανάσταση, ξεκινώντα από του μισθού, είναι καθοριστική σημασία για να εξασφαλίσουμε περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση για ολόκληρη την οικονομία. Χωρί την αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου των γυναικών, δεν θα έχουμε μια Ευρώπη ισχυρή που να μπορεί να προωθήσει τι αξίε τη. Ακόμα και στη νέα ε, ψηφιακή οικονομία, οι γυναίκε εκπροσωπούν ένα τεράστιο δυναμικό που δεν έχει αξιοποιηθεί. Ο μεγαλύτερο αριθμό των γυναικών στον τομέα τη επικοινωνία και αν ήταν μεγαλύτερο ο αριθμό αυτό, θα υπήρχε μια αύξηση 9 δι ευρώ στο ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για περισσότερη εργασία χρειαζόμαστε γυναίκε επιχειρηματίε, επαγγελματίε που να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφιακή εποχή και να έχουν απασχόληση. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική ευημερία και απασχόληση. Το να αποκλείονται από τον χώρο τη εργασία σε διεθνέ επίπεδο κοστίζει 11,5 δι ευρώ ε, και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα το 2025. Και αυτό είναι το ΑΕΠ τη Ιαπωνία, τη Γερμανία και των ΗΠΑ συνδυασμένοι. Μόνο 24% των μάνατζερ σήμερα είναι γυναίκε και 4,6% είναι, είναι υποδιευθύντριε. Ε, Επίση, 665 εκατομμύρια γυναίκε απασχολούνται λιγότερο σε σχέση με του άντρε. Αυτό γιατί είναι πολύ λίγε ακόμα γυναίκε στον τομέα των ε, τεχνολογιών, τη πληροφορία και τη επικοινωνία. Από τι γυναίκε που έχουν πτυχίο, μόνο 29 επιλέγουν αυτέ τι ε, σπουδέ και 4 να έχουν πραγματικά θέσει εργασία σε αυτό τον τομέα. Στον χώρο των μέσων μαζική ενημέρωση και των κοινωνικών δικτύων χρησιμοποιούνται ακόμα στερεότυπα για το ρόλο των γυναικών, ακόμη και με σεξουαλικό υπόβαθρο. Πολλέ φορέ, βέβαια, ακόμη υπάρχουν αντισώματα, όπω δείχνει η εκστρατεία Μητού. Υπάρχει ακόμη πολλή δρόμο που μένει να γίνει. Το Ευρωκοινοβούλιο επεξεργάζεται μηχανισμού καταγγελία για την ε, εξέταση των υποθέσεων παρενόχληση online και τη επίμονη παρενόχληση στο διαδίκτυο. Χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη ψηφιακή ε, κατάρτιση των γυναικών με ίση πρόσβαση σε θέσει εργασία. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΦΑΜ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολύτιμη εργασία τη, ε, προκειμένου να υποστηρίξει τι γυναίκε στην ψηφιακή εποχή και των χώρων των μεσομερική ενημέρωση. Επίση, Χαιρετίζω το Ευρωπαϊκό Γραβείο για του τομεί αυτού που ε, έχει προβλέψει ο Επίτροπο Γκάμπριελ. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ακόμη και ο επόμενο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβλέψει κονδύλια για την ε, μόρφωση των γυναικών και την ψηφιακή του επιχειρηματικότητα. Θα καλέσω τα κράτη-μέλη να σεβαστούν αυτέ τι δεσμεύσει στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για την ψηφιακή εποχή στο Τάλιν και για την ε, ψηφιακή εκπαίδευση με ίσε ευκαιρίε. Πολλέ αντιπαραθέσεις και πολλές καταχρήσει ξεκινούν από τον ανδρικό φόβο για τι δυνατότητε των γυναικών. Είναι ένα είδος ψυχολογικής κατωτερότητας ε, που βιώνουν οι άντρε. και αυτό πολλές φορές εκδηλώνεται με βίαιε πράξει, με περιθωριοποίηση και κατάρριξη των δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται για την ισότητα των φύλων. Δεν θα έχουμε ένα καλύτερο ε, κόσμο εάν δεν αναγνωριστεί και η αξία των γυναικών. Με δέσμευση και πάθο και στον χώρο τη εργασία. Αυτό δεν είναι μόνο μια μάχη των γυναικών για τι γυναίκε. Είναι κάτι που πρέπει να το καταφέρουμε όλοι, ε, με όλη την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Ταγιάννη, τον ευχαριστώ για αυτές τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Βέρα Γιούροβα, που είναι υπεύθυνη επίτροπος για δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Κυρία Πρόεδρε, Αγαπητοί φίλοι και συμμετέχοντες, ακούσαμε θερητικά λόγια από τον πρόεδρο Ταγιάννη και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ο πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, δεν φοβάται, δεν τον φοβίζει η δυνατότητα και οι δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες. Και αυτό είναι πολύ καλό να το ξέρουμε. Συμφωνούμε όλοι ότι η Διεθνής ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας έχει να κάνει ε, με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των γυναικών σε όλους τους τομείς. Και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ούτε στην Ευρώπη έχουμε πετύχει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχουμε κάνει πολλά, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε. Υποεκπροσωπούμεθα στην αγορά εργασίας. Δεν μπορούν πολλές γυναίκες να ακολουθήσουν το όνειρά τους, ε, τη σταδιοδρομία τους, κάτι το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματά τους. Στα μέσα ενημέρωση, στο ψηφιακό τομέα επίση υπάρχουν ακόμα πολλές διαφορές. Γι' αυτό και χαίρομαι που επιλέξατε αυτό το θέμα για τη σημερινή εκδήλωση και ευχαριστώ και την Επιτροπή Γυναικών που με κάλεσε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απ' τη μια λοιπόν η πληροφορική προσφέρει νέες δυνατότητες στην αγορά εργασίας, προσφέρει λύσεις για περισσότερη ευελιξία και ποικιλομορφία τρόπους εργασίας και συνδυασμό προσωπική και οικογενειακή ζωή. Από την άλλη μεριά όμω, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε αρκετού ειδικού στην πληροφορική, πρώτον, και δεύτερον, υποεκπροσωπείται το γυναικείο φύλλο μεταξύ αυτών. Το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Δύο Φύλων, με την έκθεσή του, λέει ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο από μία στις πέντε που έχουν δίπλωμα στην πληροφορική. Και το νούμερο αυτό δυστυχώς χειροτερεύει όσο περνάει ο καιρός. Ακόμα και οι πιο νέοι δεν ακολουθούν τέτοια σταδιοδρομία. Ακόμα και οι πιο νέες γυναίκες. Μόνο 17% των 8 εκατομμυρίων που δουλεύουν στην πληροφορική είναι γυναίκες. Και ακόμα χειρότερο υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που εγκαταλείπουν θέσεις απασχόλησης στην πληροφορική γιατί δεν μπορούν να τα συνδέσουν με άλλες ε, δραστηριότητες ή για παράδειγμα με την οικογενειακή του ζωή. Και όχι γιατί οι γυναίκες δεν έχουν τις δυνατότητες ή δεν ενδιαφέρονται. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ε, διαφορές στις δεξιότητες των νέων ανδρών και νέων γυναικών στην πληροφορική. Για παράδειγμα, το 2016 46 από ένα εκατομμύριο, μάλλον 46% ήταν γυναίκες και παιδιά σε μια μεγάλη εκδήλωση για τέτοια θέματα πληροφορικής. Δηλαδή ενδιαφέρονται οι γυναίκες, δεν ότι δεν ενδιαφέρονται. Οι διαφορές στην εκπαίδευση παίζουν σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και εκπροσωπούνται πολύ λιγότερο γυναίκες θέσεις απασχόλησης στην πληροφορική. Συνεπώς, η ενίσχυση των γυναικών ε, στον τομέα αυτό της πληροφορικής είναι κάτι που θα βοηθήσει την ισότητα. 66 στα έχουμε τώρα σαν ε, βαθμολόγηση για την ε, ισότητα σε αυτά τα θέματα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολύ περισσότερα ακόμα. Και γι' αυτό στην εντολή μου ξεκίνησα διάφορες πρωτοβουλίες που μπορούν να βοηθήσουν να υπάρξει πραγματική βελτίωση. Ένα σημαντικό θέμα που εξετάζουμε είναι ίση πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους. Δεν είναι θέμα μόνο οικονομικής ανεξαρτησίας της γυναίκας, αποτελεί και προϋπόθεση προκειμένου να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, ευημερία και ανταγωνιστικότητα. Ε, η πρόοδος δεν προχωράει αρκετά. Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στους μισθούς επιμένουν οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε ακόμα περισσότερο. Τον Νοέμβριο του 2017 ανακοινώσαμε μία απάντηση προκειμένου να μειωθούν οι διαφορές αυτές με ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο θα πρέπει να αποδώσει μέχρι τα τέλη τη εντολή μα, δηλαδή μέχρι το τέλο του 2019. Έχουμε 20 δράσεις που ανακοινώσαμε ώστε να αυξηθεί μεταξύ άλλων και η παρουσία των γυναικών στον κλάδο της πληροφορικής. Τον Απρίλιο του 2017 ανακοινώσαμε πρωτοβουλία για να βελτιώσουμε τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών στους χώρους εργασίας. Κυρίως να βελτιώσουμε τις δυνατότητες συνδυασμού της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Να φροντίσουμε να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες φύλαξης των παιδιών, φροντίδας. Επίσης να υπάρξουν οι συμμιστοί στις διάφορες επιχειρήσεις και με τους κοινωνικούς εταίρους συζητήσαμε για συγκεκριμένα μέτρα ώστε να υπάρξει καλύτερη ισορροπία και γυναικών στις θέσεις λήψη αποφάσεων. Ε, ο συνάδελφός μου, Καβριέλ. Είναι από τη Βουλγαρία, κυρία Γκάμπριελ, δεν ξέρω πω προφέρεται ακριβώ το όνομά τη, αν είναι Γκέμπριαλ ή Γκάμπριελ. Σήμερα πάντως θα παρουσιάσει με περισσότερες λεπτομέρειες αυτό το οποίο κάνει η γκαμπριελ σημερα παντω θα παρουσιασει με περισσοτερε λεπτομερειε αυτο τα οποια κανει η ευρωπαικη επιτροπη για να αντιμετωπιστεί το θέμα τη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην εκπαίδευση που όπως είπαμε είναι βασικός παράγοντας που οδηγεί στην υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις απασχόλησης στην πληροφορική. Πάντως πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε και άλλη πρόκληση που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση. Και αυτό είναι η βία online και, online και η παρενόχληση των ε, νέων ε, γυναικών, των κοριτσιών. Πρέπει να έχουμε προγράμματα στο διαδίκτυο περισσότερο ασφαλή. Δυστυχώς όλο και περισσότερα μηνύματα εμφανίζονται στο ε, διαδίκτυο, από αυτά στα 17% παρενόχλησης σε βάρος νέων κοριτσιών. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να αντιμετωπίσει ένα κορίτσι στη ζωή του τέτοια φαινόμενα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτήν την διαδικτυακή βία και σεξουαλική παρενόχληση. Χάρη στις εκστρατείες μας πάντως οι άνθρωποι παίρνουν τα ζητήματα αυτά πιο στα σοβαρά και ενθαρρύνονται τα θύματα να καταγγείλουν την βία αυτή και να ζητήσουν στήριξη. Έχουν δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και εγώ σκοπεύω να κάνω πιο εντατική ακόμα την εκστατεία μας και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξή του. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε βήμα-βήμα, προκειμένου η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων να γίνει πραγματικότητα και στον ψηφιακό κόσμο και στα μέσα ενημέρωσης. Κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσω ευχόμενοι σε εσά καρποφόρες εργασίες και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για αυτή τη Διεθνή ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας. Σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για την αδιάλειπτη συνεργασία σας και πρέπει να πω κι εγώ ότι όντως πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να υπάρξει πρόοδος τελικά στον τομέα της ισότητας των φύλων. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τώρα με χαρά σας ανακοινώνω ότι μπορώ να σας ε, παρουσιάσω δύο εξαιρετικές κυρίες, την ε, σκηνοθέτη της ε, ταινίας Le Suffragette, την κυρία Σάρα Γκαβρόν και την τραγουδίστρια και ιδρύτρια του φεστιβάλ Mad Women Fest, την κυρία Πίλαρ Χουράδο. Και έχετε το λόγο, κυρία Γκαβρόν. Καλημέρα σας. Καλημέρα αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι σκηνοθέτης, οπότε θα σας μιλήσω από αυτή την οπτική. Όλοι οι υπόλοιποι βέβαια ξέρετε πολλά περισσότερα για τα υπόλοιπα ΜΜΕ. Μου πήρε πολύ καιρό να υψώσω τη φωνή μου και τώρα που την έχω δεν πρόκειται να σταματήσω να τη χρησιμοποιώ, είπε η Μαντλίν Ολμπράιτ. Και πρέπει να πω ότι αυτός είναι, αυτό είναι το έτος που οι γυναίκες δεν σιωπούν. Βέβαια δεν, έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει πολλά αν το δει κανείς, ε, τουλάχιστον από τη δική μου οπτική, από τη βιομηχανία της ε, δημιουργίας ταινιών. Όταν εγώ τελείωσα το σχολείο, 90% ναι, των ταινιών ε, γίνονταν από άντρες. Το 2018, 90% των ε, ταινιών εξακολουθούν να γίνονται από ε, άντρες. Αλλά είμαστε ακριβώς στην χρονική στιγμή τη σωστή για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ορόσημο. Όντω πρέπει να ενισχύσουμε τι γυναίκε στα ΜΜΕ, στην τηλεόραση, στι ταινίε, γιατί οι γυναίκε αποτελούν τον καθρέφτη τη κοινωνία μα και την επηρεάζουν. Όπω και το κίνημα Time's Up είπε, τα μέσα μπορούν να παίξουν ένα τεράστιο ρόλο ώστε ο κόσμο να γίνει πιο ισότιμο. Μπορούμε να συνδέσουμε, μπορούμε να αλλάξουμε την ε, βαρύτητα και τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμο μα βλέπει. Όσο μεγάλωνα δεν καταλάβαινα ότι θα μπορούσα να έχω γίνει α, σκηνοθέτης, γιατί σε, κανένα από τα, σε καμία από τις ταινίε που έβλεπα δεν υπήρχε γυναικεία, γυναίκα σκηνοθέτης και δεν είχα κανένα α, πρότυπο. Είχα όμως ένα προσωπικό μου πρότυπο, τη μητέρα μου που ήταν εδώ σήμερα, η οποία ήταν πολιτικός βάσης και, και κατάφερε να γίνει και δήμαρχος. Και έτσι είδα την ε, επιρροή που μπορούσε η ίδια να ασκήσει. Βέβαια μου πήρε κάποιο καιρό για να καταλάβω πώς μπορούσα εγώ να καθοδηγήσω τη δική μου δύναμη και όταν ήμουν στη 20 μπόρεσα να δω ότι υπήρχαν και άλλες ε, σκηνοθέτες γυναίκες και ανακάλυψα αυτό που τώρα λέμε οι, οι μέρες των γυναικών στε, στις ταινίες. Και ήταν πραγματικά ένα σημαντικό γεγονός για να δω πώς οι γυναίκες αλλάζουν την οπτική στα ΜΜΕ η, ταινία που έκανα ήταν η ταινία που ήθελα να κάνω και φοράω και το αντίστοιχο τη ΕΡΤ όπως βλέπετε. Η ιστορία αυτή δεν είχε η υποθεί, ήταν μία από τα, ένα από τα βασικά κινήματα του 20ου αιώνα και πραγματικά ήταν έβριφε δυναμικών χαρακτήρων. Και φυσικά είχε να κάνει και με τα σύγχρονα γεγονότα στον, στην κοινωνία μας. Αλλά ο κόσμος δεν ήταν ακόμα έτοιμος για να ακούσει αυτή την ιστορία. Μίλησα με παραγωγούς ταινιών και μου είπαν ε, γυναίκες και πολιτικοί τι, τι ταινία είναι αυτή, ποιος θα τη δει. Και εγώ τους είπα γιατί να μην βάλουμε μέσα και καμιά έκρηξη, τίποτα κυνηγητά με την αστυνομία, τότε μπορεί να ενδιαφερθούν περισσότερο μου πήρε 10 χρόνια ακόμη για να ενδιαφερθεί κάποιος. Και ίσως και λόγω του ίντερνετ ξεκινήσαμε να ακούμε να μιλούν γυναίκες ε, πολύ δυνατά απέναντι στην καταπίεση, η Pussy Riot, οι άλλες ε, ακτιβίστριες και παραγωγή που μπορούσαν να υποστηρίξουν του στόχου μου. Αλλά βεβαίω τα εμπόδια ήταν πολλά για να κάνουμε την ταινία. Είχαμε πολλέ ε, ε, ηθοποιού που ήθελαν να παίξουν, αλλά έπρεπε να έχουμε και υποστηρικτικού ρόλου για άνδρε. Και υπήρχαν ατζέντιδε που διάβαζαν τα ε, τα κείμενα και μας έλεγαν «Ε, «Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλος ο ρόλος για τον ηθοποιό αυτό». «Α, καλώς ήρθατε στον κόσμο των γυναικών τα τελευταία 100 χρόνια» τους λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει καταφέραμε να προσελκύσουμε κάποιους πολύ σημαντικούς ηθοποιούς. Πολλοί εξέφρασαν την έκπληξή τους όταν άρχισαν να δουλεύουν ε, στην ταινία και μας είπαν δεν, δεν έχουν υπάρξει ποτέ ε, σε σετ που να, υπάρχει να υπάρχουν τόσα πολλά ιστρογόνα η συγγραφέα, ο σχεδιαστή, οι σκηνοθέτε, οι παραγωγό ήταν όλε γυναίκε. Ο μεγαλύτερο μύθο, μάλλον το μεγαλύτερο ψέμα, είναι ότι οι γυναίκε δεν δουλεύουν καλά μαζί. Και δουλέψαμε καλά και δουλεύουμε καλά. Υπάρχουν και άλλα βέβαια εμπόδια για το πώ πρέπει να πολεμήσει ω γυναίκα για να περάσει το μήνυμά σου και ποιε μάχε αξίζει να δοθούν. Το είδαμε και στην, ε, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ε, όταν ε, κάναμε την, το γύρισμα είπα ότι χρειαζόμαστε πρόσβαση στο Κοινοβούλιο και μας είπαν ότι δεν έχει δοθεί ποτέ άδεια για να υπάρξει γύρισμα εντό του Κοινοβουλίου, ούτε στο Mission Impossible δεν δόθηκε άδεια. Και εγώ είπα ότι πρέπει να, αρχίσουμε, να, να συνεχίσουμε να το ζητούμε μέχρι να μα τη δώσουν. Τελικά το Κοινοβούλιο είπε ναι αλλά ζήτησε περισσότερε λεπτομέρειες. Του είπα ότι θέλαμε να φέρουμε 200 ε, συμπληρωματικού ε, ε, ηθοποιούς και, και, που θα κάνουν τους αντιφρονούντες στο, στην αυλή του Κοινοβουλίου. Και θα, ως εκ του θαύματο συμφώνησαν. Οπότε μας δόθηκε πλήρης πρόσβαση στο κοινοβούλιο που ήταν ακριβώς το θεσμικό όργανο που αρνήθηκε στις γυναίκες την πρόσβαση την, τις φυλάκιζε επειδή ρωτούσαν, ε, ε, έθεταν ερωτήματα σε διάφορες πολιτικές συζητήσεις κλπ. Ήταν πραγματικά τεράστια η αλλαγή που πέτυχαν οι σουφραζέτες και μας έδειξαν ότι η αλλαγή όντως είναι δυνατή. Υπήρχε βέβαια και μια στιγμή όπου, ήταν, όπου συνεχίζει να είναι δυνατή η αλλαγή και βλέπουμε πόση μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει ένας χρόνος. Το 2017 ξεκίνησε με τις ε, διάφορες ε, διαδηλώσεις των γυναικών ε, ανά τον κόσμο και τώρα έχουμε το MeToo, το Time's Up που συνδέει τις γυναίκες σε όλους τους κλάδους και να γνωρίζουμε ότι πρέπει όντως να είμαστε συμπεριληπτικές για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το φεμινισμό χωρίς σύνορα θέλουμε και οι πιο φτωχέ γυναίκε να έχουν την ίδια αξία όσο ο πιο πλούσιο άντρα. Και θέλουμε να συνεργαστούμε και με του άντρε συμμάχου. Όλοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την υποεκπροσώπηση και την καταπίεση στα ΜΜΕ. Και ω γυναίκα σκηνοθέτη, εγώ χαίρομαι που μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για όσο χρειάζεται ώστε να έρθει η αλλαγή. Για να γυρίσω λοιπόν στη Μαντλίνο Ρομπράιτ και στα σχόλιά τη, μπορούμε να το πετύχουμε όταν δεν σιωπούμε. Και για να το προχωρήσω ακόμα παραπάνω, μπορούμε να το κάνουμε όταν ενωθούμε και όταν κάνουμε θόρυβο. Και μια που μιλάω για το να κάνουμε θόρυβο, να σας πω δύο πράγματα της Emily Pankhurst, της επικεφαλής του κινήματος των σουφραζιτών. Έχεις δύο μωρά, που είναι και τα δύο και θέλουν και τα δύο να φάνε. Το ένα είναι υπομονητικό και περιμένει όσο, όσο χρειαστεί η μαμά του για να του δώσει το φαγητό του. Το άλλο είναι ανυπόμονο και φωνάζει, κλαίει, ουρλιάζει, κλωτσάει και πραγματικά κάνει όλους να αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιο μωρό είναι αυτό που παίρνει το φαγητό του πρώτο. Αυτή ακριβώς είναι η ιστορία της πολιτικής. Πρέπει να είσαι πιο επιθετικός από όλους. Πρέπει να ε, γεμίζεις ε, το, τους ρόλους όπου υπάρχουν και πρέπει να κάνεις όσο το δυνατόν περισσότερο θόρυβο, περισσότερο από όλους τους άλλους. Οπότε όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε περισσότερο θόρυβο από οποιονδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Από βάθος καρδίας πραγματικά. Σάρα, που ήρθατε σήμερα εδώ σε αυτή την εκδήλωση. Και σας ευχαριστώ επίσης για το έργο σας, για τις δραστηριότητές σας, γιατί μέσω του δικού σας έργου αποδεικνύεται ότι οι γυναίκες σκηνοθέτες μπορούν να είναι εξίσου καλά σκηνοθέτες όπως και άντρες, γιατί όχι. Οπότε σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια του έργου σας. Επίσης χαιρετίζω και τη μητέρα σας που είπατε ότι είναι εδώ παρούσα. Τώρα θα δώσω το λόγο σε μια τραγουδίστρια που έχει οργανώσει το Matpams Festival. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία Πιλάρ Κουράδο. Καλή σας μέρα όλοι. Ευχαριστώ πολύ την Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών, την κυρία Μπλικοβιτσιούτε και την Επίτροπο Καταναλωτών Ισοδικαιωμάτων, την κυρία Γιούροβα, που με καλέσατε εδώ. Και βέβαια και την ε, συνάδελφό μου, την Σάρα Καβρών που μου δώσετε την ευκαιρία να είμαι εδώ μαζί σας. Για να συνοψίσω τι ήταν το Mad Women Fest. Οργανώθηκε επειδή οι γυναίκες αποφάσισαν να πούνε φτάνει πια. Φτάνει πια στην καταπίεση, φτάνει πια στη βία. Οι εκστρατείες όπως είναι το Too, Τσάπ και τα λοιπά, οδήγησε και στο δικό μας, που δεν είναι ακριβώς ένα φεστιβάλ, είναι μια ιδέα τουλάχιστον στο μυαλό μου ήταν έτσι, το ονειρεύτηκα ότι θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Και μέσα στο όνειρο αυτό σκέφτηκα ότι ήταν πολύ σημαντικό να μαζέψουμε τις γυναίκες που αριστεύουν στις τέχνες. Γιατί συνήθως βλέπουμε πρότυπα που μας κάνουν να λέμε ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως θα θέλαμε. Οι γυναίκες μένουν έξω από το σύστημα. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτές οι εξαίρετες γυναίκες αυτές που είναι σε θέση να ονειρευτούν ένα διαφορετικό κόσμο, να δημιουργήσουν ένα, άλλο σύμπαν και αυτές οι γυναίκες θα έπρεπε να μπορούν να έχουν αρκετά, να εξοπλιστούν αρκετά από την κοινωνία ώστε να μπορέσουν να κάνουν ε, το όραμά τους πραγματικότητα. Και εμείς αυτό θέλουμε. Όλες οι γυναίκες των τεχνών και αυτές να επωφεληθούν και να δείξουν στον κόσμο ότι τα πράγματα μπορούν να είναι διαφορετικά, ότι μπορούμε να τα κάνουμε αλλιώς και πάνω απ' όλα ότι μπορούμε να δείξουμε την συνέστησή μας απέναντι στους άλλους και όλοι μαζί να βρούμε ένα νόημα και το όνειρό μας να γίνει κανονικότητα. Αυτό προσπάθησε να κάνει και το Mad Woman Fest. Δεν βέβαια μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε και τους άντρες. Γι' αυτό εδώ δεν ήρθα μόνο για να σας παρουσιάσω τις γυναίκες αυτές των τεχνών, αλλά ήρθα για να ζητήσω και τη στήριξη των ανδρών και να σας πω ότι υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν στην ισότητα και που θέλουν και αυτοί και πιστεύουν σε έναν άλλο κόσμο. Έτσι και αυτοί δέχτηκαν ονομαστούν Mad Woman. Τι είναι Mad Woman είναι οποιοδήποτε έχει την τρέλα να μπορεί να δει πιο μακριά και να πιστέψει σε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω όλοι εσείς λοιπόν να το δεχτείτε και να γίνετε κι εσείς Mad Woman μαζί μας. Θέλω επίσης να, να σας πω ότι όταν μιλάμε για την εκπροσώπηση των γυναικών, ο μόνος τρόπος είναι να επιτρέψουμε σε όσο γίνεται περισσότερες γυναίκες να δείξουν τι μπορούν να κάνουν, να δείξουν τις δεξιότητές τους, τα ταλέντα τους. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Κάθε μία όμως από αυτές τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ή γενικά εκδηλώσεις που δώσαν φωνή στις γυναίκες αυτές ήταν ακριβώς για να δώσουν φωνή σε αυτές που δεν την είχαν αυτή τη φωνή. Στις περιπτώσεις αυτές που δεν μπορούσαν να ακουστούν οι γυναίκες. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν αγγίξεις τον άλλο στην καρδιά του, πολύ πιο εύκολα θα το κάνεις να καταλάβει τι νιώθεις. Πρέπει η ενσυναίσθηση αυτή να περισχύσει, να μας κάνει να μπορούμε να δούμε τον κόσμο και με τα μάτια του άλλου. Ο κόσμος αυτός λοιπόν της τεχνολογίας, ο ψηφιακός, που δείχνει, μας κάνει μάλλον να νομίζουμε ότι έχουμε πρόσβαση στα πάντα, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ότι τελικά οδηγεί στα ίδια ασφάλματα που έχουμε οδηγηθεί όλα αυτά τα χρόνια στην κοινωνία μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε τα πράγματα τώρα αλλιώς και να δώσουμε πρόσβαση στον νέο αυτό κόσμο σε όλες τις γυναίκες και σε όλο τον κόσμο. Να νιώσει ότι αυτές οι ευκαιρίες ε, δεν θα πέσουν στις ίδιες παγίδες ε, της καταπίεσης που είχαμε στο παρελθόν. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, που κάνουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, μου εξήγησαν πόσο πολύ δυσκολεύονται να κάνουν τη δουλειά του. Γιατί, γιατί είτε από το πανεπιστήμιο, από τη σχολή του νιώθουν την καταπίεση των γυναικών σε βάρο τους. Ο μόνο τρόπο λοιπόν για να πετύχουμε είναι να φροντίσουμε και οι άλλοι να αποτελέσουν μέρο τη δικιά μα τη ζωή και εμεί να αποτελέσουμε μέρο τη ζωή των άλλων. Εμεί είμαστε οι άλλοι και οι άλλοι είμαστε εμεί. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στον κόσμο της ψηφιοποίησης που έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κλείνονται ε, μέσα σε έναν ε, πολύ περιορισμένο χώρο και να ζουν μια διαφορετική ζωή από τη δικιά τους. Την πρώτη όπερα που συμμετείχα εγώ, την είχε γράψει μια γυναίκα στο Τεάτρο Ρεάλ το 2011 στη Μαδρίτη και έπρεπε να περιμένουμε μέχρι το 2011 ώστε μια γυναίκα να ανεβάσει μια όπερα στο Τεάτρο Ρεάλ της Μαδρίτης. Λοιπόν, γίνονται πράγματα, ανοίγουν πόρτες, αλλά σήμερα συμβαίνει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είναι ότι πάρα πολλές γυναίκες στον κόσμο αποφάσισαν να πούνε σήμερα ότι ναι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα της καινούργια μας ζωής. Της ζωής όπου ο κόσμος θα αλλάξει. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό και να το κάνουμε πραγματικότητα. Θέλω επίσης να διεκδικήσω από όλες τις γυναίκες που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και που δεν θέλουν να είναι ουτοπία η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ε, να ξέρουν ότι μερικές φορές πρέπει να πληρώσουμε ένα υψηλό τίμημα. Για πολλές ε, έχει γίνει πραγματικότητα αυτό. Άλλες πριν όμως χρειάστηκε να πληρώσουν ιδιαίτερα ψηλό τίμημα. Για μένα η Πιλάρ του Βινιάνια που είναι Μία γυναίκα που έχασε τη ζωή της παλεύοντας για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Ισπανία, τη δικτατορία. Ήταν στην αντίσταση και έκανε πάρα πολλά για να ενώσει τον κόσμο υπέρ της ελευθερίας. Η γυναίκα αυτή ήταν μια γυναίκα που, τι ξέρω το όνομά της δηλαδή, ξέρω, ήταν ε, προγιαγιά μου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να διεκδικήσουμε αυτή την ιστορική μνήμη γιατί είναι ο σωστός τρόπος να πούμε στον κόσμο ότι δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Επίσης θέλω να σας πω ότι για το φεστιβάλ αυτό, το Mad Woman Fest, να ξέρετε ότι δεν θέλουμε να είναι ένα φεστιβάλ μόνο της Ισπανίας, θέλουμε να είναι παγκόσμιο, στον κόσμο ολόκληρο. Ήδη με την πρώτη του έκδοση κινητοποιήθηκε ακόμα και η Ισπανική κυβέρνηση και ο και πήραμε βραβεία. Και τώρα βρίσκομαι και εδώ, μαζί σας. Θέλω λοιπόν να είναι κάτι ευρωπαϊκό επίσης και να ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι που ανήκει στην Ευρώπη. Αυτό είναι η τέχνη που είναι δύναμη. Και αυτή η δύναμη που ζητάτε για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες περνάει μέσα από τη δύναμη της τέχνης. Δεν το ξέρετε, αλλά θέλω εδώ να σας πω, να ανακοινώσω ότι φέτος θέλω να βραβεύσω δύο εξαίρετους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Την πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών, την κυρία Βικεβιτσιούτε πρώτα απ' όλα, να τη βραβεύσω στο φεστιβάλ αυτό και την κυρία Γιούροβα. Θέλω να είσαστε τα δύο βραβεία του Mad Women Festival του 2018. Και αυτό γιατί το έργο σας για τις γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί υπάρχουν πράγματα όπως η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που είναι κάτι εξαιρετικό και που έχει προωθήσει η κυρία Γιούροβα. Θα έπρεπε λοιπόν να αναγνωριστούν όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Ελπίζω θα είμαστε στο Βερολίνο φέτος, αλλά ελπίζω κάθε χρόνο να καταφέρνουμε μία διαφορετική χώρα ευρωπαϊκή να προσκαλεί το φεστιβάλ αυτό και έτσι να κυκλοφορήσουμε σε όλη την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη τι είναι, είναι η Ευρώπη της ελευθερίας, της ποικιλομορφία ανδρών και γυναικών που αγωνίζονται και συνεχίζουν να αγωνίζονται ώστε ο παλιός αυτός κόσμος να αλλάξει και να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για το μέλλον. Τι άλλο να σας πω, σίγουρα πολλά θα μπορούσα να σας πω, αλλά ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πολλοί μου ζήτησαν να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω καλύτερα, να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να τραγουδήσω, τέλος πάντων θα χρησιμοποιήσω, παρόλο που δεν ξέρω πόσο σχέση έχει, αν και μπορεί και να έχει. Ρωσίνη, είναι τα 100 χρόνια του Ρωσίνη. Το έχω τραγουδήσει πολλές φορές. Τη Ρωσίνα. που συμβολίζει τη δύναμη των γυναικών. Προκειμένου ο κόσμος να γίνει όπως θα έπρεπε να είναι. Ο κόσμος αυτός μας ανήκει σε όλους μας. Αυτό. Επιτρέψτε μου λοιπόν, μια στιγμή μόνο, για να σας χαρίσω τη φωνή μου, ευχαριστώντας σας για όλα έχετε κάνει για μας. Ξεκινάει μια πρωτοβουλία για να κουνηθεί ο κόσμος, να αλλάξει. Εσείς κάνετε τους νόμους γι' αυτό όμως. Ταρά σας από τα βάθη της καρδιάς μου σας συγχαίρω. Κυρία Χουράδο, δείξατε το ταλέντο σας, το χάρισμά σας και αυτή την τεράστια δύναμη που έχουν οι γυναίκες. Τη δύναμη να εκφραστούν με την τέχνη. Μια δύναμη που μπορεί να μας φέρει κοντά, που να μας επιτρέψει να κάνουμε τις ίσες ευκαιρίες πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά. Σας εύχομαι κάθε τύχη για τα φεστιβάλ σας και ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να ταξιδεύετε στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για να ε, μεταδίδετε αυτές τις αξίες και τα ιδανικά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα συνάδελφοι. Θα ευχαριστήσω όλες τις μετέχουσες ε, στο αρχικό πάνελ, την Επίτροπο, την σκηνοθέτηδα, την τραγουδίστριά μας. Ε, το πρώτο μέρος αυτής της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε και τώρα θα προχωρήσουμε στις συζητήσεις που είναι οργανωμένες σε πάνελ. Θα παραδώσω την Προεδρία στις ε, διευθύντριες του πάνελ που θα διευθύνουν τη συζήτηση στις συντονίστρες. Την ε, κυρία Ροντρίγκης λοιπόν προσκαλώ στην, ε, στο Προεδρείο. Την κυρία Γκιουλσούν Μπιλγκεχάν, η οποία είναι από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και την κυρία Μικαέλα Σόιντροβα, που είναι Ευρωβουλευτής. Τα τρία σημερινά πάνελ θα ασχοληθούν με τα εξή θέματα. Η διαμόρφωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, και γυναίκες, η χειραφέτες των γυναικών μέσω της ψηφιακής ε, ε, ενδυνάμωσης και οι γυναίκες και τα κορίτσια στην ψηφιακή εποχή. Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για να πάρουν τη θέση τους ομιλήτριες στο πάνελ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο πάνελ. Έχουμε την τιμή να έχουμε στο πάνελ αυτό την κυρία Γκυλσούν Μπίλγεθαν, μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και την κυρία Μικαέλα Σόιντροβα, Ευρωβουλευτή και υπεύθυνη συγκήτρια για, το, για την έκθεση Ισότητα των Φίλων στον τομέα των μέσων μαζική ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα περάσω τώρα στη μητρική μου, την Πορτογαλική. Το να δημιουργήσουμε κοινωνίε ίσων ευκαιριών είναι προτεραιότητα των σύγχρονων κρατών. Υπό αυτήν την έννοια, όλη η επικοινωνιακή μας πολιτική θα πρέπει να αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο στο να οικοδομήσουμε μια κοινωνία όπου άντρες και γυναίκες μπορούν να έχουν ίσα δικαιώματα. Θα πρέπει να προωθήσουμε και να επιταχύνουμε τις ε, ε, εξελισσόμενες μεταρρυθμίσεις και να φροντίσουμε την εφαρμογή τους πέραν των κατακτήσεων που τώρα έχουμε πετύχει, ακόμη παραμένουν στερεότυπα και διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών. Η θέση ανδρών και γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι ίση. Οι άνδρες καθορίζουν τα πράγματα. Επίσης υπάρχει η ελληπής εκπροσώπηση των γυναικών στον χώρο των κοινωνικών ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης εκεί όπου υπάρχουν ε, λήψεις και εκεί όπου λείπει εμπειρογνωμοσύνη για να αναλάβουν το ρόλο που τους αρμόζει. Θα πρέπει επίσης να καταγράψουμε εδώ ότι στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων και της επικοινωνίας έχουμε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Το πρώτο βήμα είναι να το εντοπίσουμε και το δεύτερο να φροντίσουμε το περιεχόμενο με μία προοπτική των δύο φύλων να επιτρέψει μια αποτελεσματικότερη έκφραση στις γυναίκες. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα πρέπει να αρχίσει να υπάρχει και μια θετική ε, διακριτική μεταχείριση, μεταβατικού χαρακτήρα. Αν όμως θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα με τρόπο προοδευτικό, πρέπει όλοι να αναλάβουν το ρόλο τους. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε το σύστημα της ισότητας του φύλου και της πρόθεσής του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας κανόνες και πρότυπα σε σχέση με την επαγγελματική σταδιοδρομία και την ε, ε, έκφραση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ίδιο και με προστασία και με τις ανάλογες ε, κυρώσεις. Το ίδιο και στην εκπαίδευση και με την ε, διαμόρφωση ενεργών πολιτικών για τον συνδυασμό επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και για την καταπολέμηση των ε, ηθικών και συστικών στερεοτύπων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει επίσης ο αλφαβητισμός και η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας να καλλιεργηθεί περισσότερο. Θα πρέπει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να προωθήσουμε αυτή την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς στις κοινωνίες μας. Και το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει τη δική του ευθύνη για την επίταξη αυτού του στόχου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν προχωρήσουμε, θα περάσω τώρα στα αγγλικά. Θέλω να σας παρουσιάσω κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να είναι διαδραστική η συζήτησή μας και να ζωντανέψει λίγο. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι μπορείτε να αποστάρετε την εκδήλωση αυτή στο Twitter με το hashtag IWD2018. Έπειτα, να σας ενημερώσω ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο που ονομάζεται Slido. Έτσι, Σλάιντο, έτσι, ναι. Ε, δεν ήμουν σίγουρο αν ήταν σλάιντο ή σλίντο. Για να μπορεί το κοινό να απαντήσει σε γκάλοπ και να θέσει ερωτήματα κατά την ε, ε, εξαγωγή των πάνελ Ερωτήσεις που μπορεί να θέσουν και οι πανελίστοι ίδιοι, αν έχουμε χρόνο. Εάν έχετε ένα smartphone, ένα tablet ή laptop, αρκεί να κάνετε logon στο, slide, ε, στο slide.do και να βάλετε τον κωδικό της εκδήλωσης IWD 2018. Θα σταματήσω για λίγα δευτερόλεπτα για να μπορέσετε να ανοίξετε την εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή, παρακαλώ. Okay. Εντάξει. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στο κοινό επιτρέπει στο κοινό να απαντάει σε ερωτήσεις για τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Στην αρχή του κάθε πάνελ θα ενεργοποιούμε αυτό το εντό εισαγωγικών γκάλωπ με ερωτήσεις που θα μπορείτε να απαντήσετε σχετικά με το θέμα του κάθε πάνελ. Και στο τέλος ο συντονιστής ή η η θα δίνει τις απαντήσεις που προέκυψαν από τη συλλογή των απαντήσεων. Ας ε, δοκιμάσουμε τώρα με δύο δοκιμές, δύο πειράματα. Η πρώτη ερώτηση είναι, από ποια χώρα είστε. Ανοιχτή ερώτηση, μπορείτε να γράψετε τη χώρα που θέλετε. Σας δίνω 10 δευτερόλεπτα. Όπως βλέπετε, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο World Cloud. Και βλέπετε από πόσες διαφορετικές χώρες είναι ο κόσμος που βρίσκεται σήμερα στην αίθουσα. Δεύτερη ερώτηση, δεύτερο γκάλωπ. Από ποιο φορέα ή θεσμικό όργανο είστε. Είναι multiple choice η ερώτηση, μπορείτε να, οι απαντήσεις δηλαδή, μπορείτε να διαλέξετε από τις απαντήσεις που σας διατίθενται. περισσότεροι από ό,τι θέλετε είμαστε από το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι περίεργο. Όπως βλέπετε τα αποτελέσματα είναι στην οθόνη. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στο κοινό να θέσει και ερωτήματα προ του συμμετέχοντε στο πάνελ. Θα ήθελα να θυμίσω ότι τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωβουλευτέ μπορούν απλώ να υψώσουν τα χέρια του ή να συμπληρώσουν και τις ε, καρτέλες για να ζητήσουν το λόγο όπως έχουν μοιραστεί στην αίθουσα. Ε, όσοι είναι μέρος του κοινού και δεν μπορούν να παρέμβουν στη συζήτηση διαφορετικά, μπορούν να συμβάλλουν μέσω του εργαλείου αυτού. Θα σας ζητήσω να κάνετε ένα κλικ στο συμβολάκι thumbs up, στο πλευρό αυτή τη εφαρμογή. Οι πιο δημοφιλεί ερωτήσει, ανάλογω με το πόσε ψήφου πάρουν, θα τεθούν στου ε, συμμετέχοντε στο πάνελ, αν έχουμε αρκετό χρόνο. Δύο ερωτήσεις δείγματα στην οθόνη. Πρώτα απ' όλα, πώς νομίζετε ότι πρέπει να απεικονίζονται οι γυναίκες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η δεύτερη, πώς νομίζετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες. Μπορείτε να ψηφίσετε την ερώτηση που προτιμάτε ή να θέσετε μια διαφορετική. I do hope you will enjoy using this tool for our events. Ελπίζω να σας ευχαριστήσει αυτό το εργαλείο και να βοηθήσει τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Για το, δεύτερο, για το πρώτο πάνελ έχουμε δύο ε, γκάλοπ. Εάν θέλετε συμμετέχετε στην, ε, ε, στις απαντήσεις και θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος. Η πρώτη ερώτηση είναι ποιο είναι το ποσοστό των ε, ε, υποθέσεων και ιστοριών που κατέγγειλαν οι γυναίκε στα μέσα μαζική ενημέρωση στον κόσμο το 2015. Πρώτα απ' όλα 13%, μετά 37% και μετά 65%. Δεύτερο, ποιο νομίζετε ότι είναι το ποσοστό γυναικείων χαρακτήρων σε ταινίες στα πρώτα 100 ε, φιλμ και ταινίες ε, φαντασίας ε, και αφήγησης το 2016 στην Αμερικανική αγορά με προκλητική ένδυση. Τα ποσοστά είναι 10,9%, 25,9% και 50,7%. Εάν το κοινό ή όσοι παρακολουθούν από το web streaming την εκδήλωση έχουν κάποια ερώτηση προς την κυρία Μπιλγκεχάν, παρακαλώ γράψτε την ερώτηση στο slide.do ή ψηφίστε για την ερώτηση που προτιμάτε και η κυρία Μπιλγκεχάν θα προσπαθήσει να απαντήσει τις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις του κοινού. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκυλσούν Μπιλγκεχάν. Με συγχωρείτε με την πορτογαλική μου προφορά, δύσκολα από σωστά το όνομά σα, μέλο τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Περίπου 7 λεπτά. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, 8 Μαρτίου, μια μέρα σημαντική για τις γυναίκες. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που βλέπω ότι μια τόσο ωραία και δυνατή φωνή ε, ακούστηκε σε αυτή την αίθουσα. Η κυρία Χουράδο νομίζω ήταν μια υπέροχη φωνή για να ξεκινήσει με την ημέρα. Την ευχαριστώ λοιπόν και τη συγχαίρω. Συνάδελφοι, κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, για σας όλους και όλες, είναι μια αφορμή για να σκεφτούμε ότι άλλο ένα έτος πέρασε και ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει ένας στόχος που δεν έχει επιτευχθεί. Ο τίτλος της παρουσίασής μου σήμερα θα έπρεπε να είναι οι γυναίκες διαμορφώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι γυναίκες τους δίνουν σχήμα και μορφή. Όμως η ερώτηση τίθεται και αυθορμήτως. Είναι πραγματικά οι γυναίκες αυτές που διαμορφώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μήπω είναι απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαμορφώνουν τις γυναίκες και το ρόλο τους. Είναι δύο ερωτήσεις στις οποίες δυστυχώς γνωρίζουμε τις απαντήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή 47 χώρες, οι γυναίκες είναι ξεκάθαρα ε, λιγότερο εκπροσωπούμενες σε όλα τα επίπεδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερως ό,τι αφορά τις θέσεις ευθύνη και το επίπεδο λήψης αποφάσεων. Αυτό που εμποδίζει την πρόοδό του σε όλου του τομεί τη οικονομία είναι αυτό που τι εμποδίζει και σε αυτόν τον κλάδο. Παρ' όλα αυτά είναι παρούσε ε, στην καθημερινότητα των μέσων μαζική ενημέρωση και στι ζώνε πολέμου και ανθρωπιστικών κρίσεων. Το γνωρίζω αυτό διότι είμαι μητέρα δημοσιογράφου. Η κόρη μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Συρία. Ανησυχώ για τη ζωή τη, είναι η μαμά τη, αλλά ταυτόχρονα είμαι και περήφανη, διότι είναι μια δημοσιογράφος, γυναίκα, τολμηρή, αγαπάει τη δουλειά τη και αναλαμβάνει του κινδύνους που χρειάζεται για να ασκεί τη δημοσιογραφία. Να πω ότι υπάρχουν και άλλε γυναίκε δημοσιογράφοι σε άλλου τομεί, όπω τον τομέα τη ερευνητική δημοσιογραφία, που πολλέ φορέ ε, διακινδυνεύουν την ίδια του τη ζωή, Όπω το είδαμε στην περίπτωση τη δολοφονία τη δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα στη Μάλτα. Εκεί όπου θα έπρεπε να γίνουν όλε απαραίτητε έρευνε για να φωτιστεί η υπόθεση. Οι γυναίκε που εργάζονται στα μέσα μαζική ενημέρωση δεν διαφεύγουν από την άδικη πραγματικότητα τη μισθολογική διάκριση μεταξύ των δύο φύλων. Για ίση δουλειά πληρώνονται λιγότερα από ό,τι οι άντρε συνάδελφοί του. Αυτό φάνηκε και από την αρχισυντάκτρια του BBC της Κέρι Γκέισι που πρόσφατα ε, από τα καθήκοντά της μετά από 30 χρόνια για να καταγγείλει αυτή τη μισθολογική κουλτούρα μέσα στην αδιαφάνεια και την παρανομία, ακόμη και στο επίπεδο της κρατικής ε, ε, βρετανικής τηλεόρασης. Χάρη σε αυτήν την χειρονομία, οι γυναίκες βρέθηκαν στα πρωτοσέλιδα. Μετά την ε, ε, έκθεση της συναδέλφου μου από την Γερμανία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Ελβίρα Γκρέις, για, για την κατάσταση των δημοσιογράφων γυναικών στην Ευρώπη και τον μισθό τους. Εκείνες κερδίζουν 16% λιγότερο από ό,τι άντρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χάσμα αυτό φτάνει και το 24% στο Βέλγιο από ό,τι μαθαίνουμε. Εκεί μόνο 30 γυναίκες δημοσιογράφοι υπάρχουν και το ποσοστό είναι ε, κανονικά 45% των γυναικών. Οι γυναίκες εγκαταλείπουν το επάγγελμα αυτό ή αποφεύγουν ακόμα και να το ξεκινήσουν επειδή είναι επισφαλής η κατάστασή τους και η θέση τους. Λιγότερο απασχολούνται σε θέσεις πλήρους ε, ε, εργασίας και πολλές φορές βρίσκονται σε θέσεις επισφαλής. Οι σταδιοδρομίες των γυναικών είναι πιο βραχίες από ό,τι των ανδρών και συνήθω οι απουσίε του είναι περισσότερε από των ανδρών επειδή έχουν και τα παιδιά. Το να ασκεί κανεί τα γονέκα του καθήκοντα ενώ είναι και δημοσιογράφο είναι αρκετά δύσκολο. Ακόμη πιο πολύ ισχύει αυτό διότι ζούμε στην ψηφιακή εποχή και η μέρα εργασία δεν τελειώνει με την σύνταξη ή την αρχισυνταξία αλλά συνεχίζεται και στο σπίτι είναι ένα φαινόμενο που διαρκώς διωγγώνεται. Οι γυναίκες δημοσιογράφοι είναι ευάλωτες ε, επίσης είναι και θύματα της παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Και οι άντρες είναι θύματα, αλλά οι γυναίκες, ιδίως αυτές κάτω των 30 ετών, συνήθως ε, είναι θύματα παρενόχλησης με ισογενικές αποχρώσεις, με σεξιστικά στερεότυπα στο χώρο εργασίας τους, κάτι που αναγκάζει τις γυναίκες που εργαζόνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ανέχονται φαινόμενα σωματικής βίας. Οι Μισέ γυναίκες έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και ε, τα τρία τέταρτα ε, εκφοβισμό ή ε, πιέσεις. Είναι ε, σαφές ότι ο ρόλος των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακριβώς εκφράζει την ανισότητα των δύο φύλων και την ευρεία διάδοση στερεοτύπων και προκαταλήψεων που ακόμη ε, εμένουν στις κοινωνίες μας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πολλαπλασιάζουν και τα προβάλλουν ακόμη περισσότερο στην ε, σκέψη των ανθρώπων. Οι γυναίκες είναι λιγότερο προβεβλημένες από τους άντρες και όταν προβάλλονται συνήθως αναλαμβάνουν παραδοσιακούς ρόλους και εκτιμώνται για προσόντα όπως η ομορφιά τους, η γλυκύτητα του χαρακτήρος, η ικανότητά τους να τα συγχωρούν όλα, ακόμα και την βία εις βάρος τους. Έχουμε όλες αυτές τις αρετές, αλλά έχουμε και άλλες, και άλλα χαρακτηριστικά πέραν αυτών. Δεν είναι τυχαίο που η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ε, που αναφέραμε προηγουμένως, ε, το πληρέστερο εργαλείο παγκοσμίω και έχει συντάξει το Συμβούλιο της Ευρώπης, και που εσείς οι ίδιοι στο Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνατε και υπογράψατε πρόσφατα, δεν είναι τυχαίο που η σύμβαση αυτή έχει σκοπό να προλαμβάνει και να καταπολεμά τη βία εις βάρος των γυναικών με συγκεκριμένες διατάξεις για το ρόλο του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, προσπογράφοντας τη σύμβαση αυτή, τα συμβαλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενθαρρύνουν τους φορείς του ιδιωτικού τομέα και τους ε, φορείς των, κοινωνιών, των ε, εταιριών της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωση να σεβαστούν την ελευθερία της έκφρασης και την ανεξαρτησία των γυναικών, συμμετέχοντας στην χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών, καθώς και κατευθυντηρίων γραμμών και προδιαγραφών αυτορύθμισης, ώστε να προλαμβάνεται η βία εις βάρος των γυναικών και να ενισχυθεί ο σεβασμός της αξιοπρέπειάς τους. Είμαι ταυτόχρονα και βουλευτής από την Τουρκία, μια χώρα όπου το επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι πραγματικά πολύ δύσκολο στην άσκησή του. Αλλά θα ήθελα εδώ να παραθέσω και μια άλλη ομάδα, την ομάδα Ντουάν, ε, που την διευθύνει τέσσερις γυναίκες οι οποίες είναι ιδιαίτερα ενεργές και έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία εδώ και χρόνια για να καταπολεμήσουν την βία ακριβώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να επιστοποιήσουν το κοινό. Έχουν δημιουργήσει και μια ειδική τηλεφωνική γραμμή που δέχεται κλήσεις για τα θύματα βίων ε, συμπεριφορών. Ε, επεισοδίων. Αυτό έχει επιτρέψει την ευαισθητοποίηση και την μεγαλύτερη κατανόηση αυτού του προβλήματο. Επίση, θέλω να δώσω και ένα παράδειγμα από την Ισλανδία. Μία από τι χώρε με την περισσότερη ισότητα στον κόσμο. Ε, υπάρχει Διεθνή ημέρα των γυναικών για τα μέσα μαζική ενημέρωση από το 2016. Με στόχο να αντιμετωπιστεί η ελληπή εκπροσώπησή του στον χώρο αυτό με μία μέρα σύμβολο. Η ε, επίσημη αλυσί, το επίσημο κανάλι ραδιοφώνου και τηλεόρασης της Ισλανδίας ε, απασχολεί 38 γυναίκες και με 38% γυναίκες και 52% άντρες στο σύνολο των εργαζομένων. Από το 2016 αποφάσισαν να αλλάξουν ε, αυτό το ποσοστό ε, ως παράδειγμα για να ακολουθήσουν και άλλες χώρες για τα μέσα μαζική ενημέρωση στο διαδίκτυο έχουμε ένα άλλο μέτωπο για τη μάχη τη ισότητα των φύλων μεταξύ και γυναικών. Εκεί υπάρχουν πολλέ φορέ εξιστικέ εκφράσει ή εκφράσει μίσου ει βάρο των γυναικών και ιδίω των πολιτικών, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτε. Ε, ακόμη πιο εύκολα στο διαδίκτυο. Μπορεί να υπάρχουν περιεχόμενα ε, προσβλητικά ή με σεξιστικό, σεξουαλικό χαρακτήρα. Η τεχνητή ευθεία η ίδια να παράγει τα ε, στερεότυπα της κοινωνίας μας, δηλαδή και το σεξισμό. Και αυτό για να αντιστρέψουμε αυτήν την τάση θα πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των γυναικών και κοριτσιών στον τομέα των επιστημών και των τεχνολογιών της ε, επικοινωνία και της πληροφορικής. Θα πρέπει να μην υπάρξει ψηφιακό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αυτό να το δούμε και στις μελλοντικέ προοπτικές της ισότητας των φύλων και των αποτελεσμάτων που θέλουμε να πετύχουμε. Κυρία, και, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για να εξαλειφθεί η διακριτική μεταχείριση και να εγκαθιδρυθεί η ισότητα. Χρειάζεται μια ε, σειρά από που έχουν σωστά εντοπιστεί στις εκθέσει, τις συστάσεις και τα ψηφίσματα των οργάνων και των ε, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το ίδιο και στα νομοσχέδια και τα προγράμματα δράσης ε, των κρατών μελών. Πρέπει όμως να εφαρμοστούν. Η χώρα με Τουρκία ήταν η πρώτη που υπέγραψε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά αν δούμε τι αποτελέσματα επετέφθησαν, δεν αρκεί κανείς να υπογράφει και να κυρώνει, πρέπει και να εφαρμόζει. Πέρασε λοιπόν μια ακόμα χρονιά και η ισότητα ανδρών και γυναικών παραμένει ένα πιαστό όνειρο. Θα πρέπει λοιπόν να ε, βεβαιωθούμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, ω απαραίτητο σύμμαχο θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου. Ίσως είδατε την ταινία The Post που αφηγείται την καθημερινότητα της Washington Post όπου μια γυναίκα, μια τολμηρή γυναίκα που δεν είχε δουλειά μπόρεσε να συνεχίσει ε, την ε, ε, έκδοση της εφημερίδας της παρά τις πολιτικές πιέσεις. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που θα μπορούσαμε όλοι να ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια σας. Και τώρα 20 λεπτά συζήτηση διότι έχουμε ήδη καθυστερήσει. από την Ουγγαρία. Μάρτα Ματράη από την Εθνική Βουλή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, γιατί οι ε, ειδικοί ανάπτυξη της ψυχολογίας λένε ότι τα ΜΜΕ επηρεάζουν την πνευματική και ψυχική υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι διαφημίσεις, τα πλακάτ, μας γεμίζουν με πληροφορίες και αυτό έχει διάφορες επιρροές στους ανθρώπους. Το περιβάλλον των ΜΜΕ βεβαίως ε, καθημερινώς αλλάζει και κυρίως αυτοί που επηρεάζονται πολύ είναι οι νέοι. Τα ΜΜΕ μπορούν να επηρεάσουν τις απόψεις τους. Και η χρήση βεβαίω των, ε, των μέσων κοινωνική δικτύωση μπορεί να οδηγήσει σε πνευματικέ ασθένειε. Το 2016 η Ουγγαρία ξεκίνησε μια ψηφιακή στρατηγική για την προστασία του παιδιού με, τη, με ενισχυμένες προτεραιότητες για, την, για μέτρα για την προστασία ακριβώ των παιδιών. Οι εθνικές αρχές για τα μέσα και το ραδιόφωνο που έχουν ε, πρόεδρο γυναίκα ε, εξέδωσαν μία έκθεση για την εκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της τηλεόρασης. Και διαπιστώθηκε ότι στα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης οι γυναίκες ε, παρουσιάζονται μέσα στα πλαίσια των ε, στερεοτύπων που υπάρχουν. Το 2017 το ποσοστό των γυναικών στις, ε, στη δημόσια τηλεόραση ήταν 24%. Η εκπροσώπηση των γυναικών σε όλη την Ευρώπη δυστυχώ είναι αρκετά χαμηλή. Οι γυναίκε είναι σε θέση να φέρουν μια θετική αλλαγή στα ΜΜΕ και μπορεί, μπορούμε επίση να δούμε ότι χρειαζόμαστε ισχυρέ οικογένειε, ισχυρέ κοινωνίε και ένα ισχυρό κράτο μπορεί να χτιστεί μόνο με ισχυρέ οικογένειε. και αυτό σημαίνει πνευματική, ψυχική, σωματική προστασία οι γυναίκες λοιπόν μπορούν να κάνουν την αλλαγή αυτή, κυρίως ε, βεβαίως όταν οι γυναίκες ζουν σε μια χώρα που δίνει έμφαση στις οικογένειες και στην υποστήριξη των οικογενειών, των παιδιών, σε μια υγιή κοινωνική πολιτική, σε μια υγιή οικονομική πολιτική, σε μια εξασφαλισμένη ηλικία συνταξιοδότησης και όταν δημιουργούνται θρησκευτικέ και κοινωνικέ ομάδε. Ε, αλλά βεβαίω αυτό μόνο με του άντρε μαζί μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μόνο μαζί με του άντρε θα είναι πλήρε οι κοινωνίε. Ευχαριστώ. Ε, ε, ναι, μου γίνονται παράπονα. Μου ζητούν οι διερμηνεί να μιλάτε αν γίνεται λίγο πιο σιγά για να σας προλαβαίνουμε. Από την Κύπρο η κυρία Αριστίδου, συγγνώμη για την προφορά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι κατεξοχήν ανταγωνιστικός. Η υφιστάμενη εργασιακή κουλτούρα και περιβάλλον αναπαράγουν τα κυρίαρχα αντρικά πρότυπα, δυσχεραίνοντας τη γυναική εκπροσώπηση στο εργατικό δυναμικό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας που έγιναν δυστυχώς για την Κύπρο είναι απογοητευτικά. Το ποσοστό της παρουσίασης των γυναικών στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τις εφημερίδες ανέρχεται στο σε 19%, ενώ στο Twitter και το ίντερνετ είναι μικρότερο από 7%. Στου τομεί τη πολιτική και τη διακυβέρνηση, η παρουσία των γυναικών ανέρχεται σε 30%. Στι ειδήσει κυριαρχούν οι άντρε δημοσιογράφοι με ποσοστό 88%, ενώ στην τηλεόραση 46% των παρουσιαστών είναι γυναίκε. Στην περίπτωση τη Κύπρου, τονίζεται η ανάγκη προβολή περισσότερων γυναικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα που μονοπολούν στι ειδήσει, όπω για παράδειγμα η οικονομία και το κυπριακό πρόβλημα. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη επένδυσης επαρκών οικονομικών πόρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα απευθύνονται σε επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πρακτικές τους, την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους σε θέματα ισότητας ώστε να καταπολεμηθεί ο σεξισμός στη γλώσσα και να επιτευχθεί πιο ισορροπή και απαλλαγμένη από στερεότυπα απεικόνηση των φύλων στι ειδήσει. Η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματο, ώστε να καλλιεργεί τι αρχές της ισότητα είναι υψή τη σημασία. Θα πρέπει επίση να υλοποιηθούν μέτρα θετική δράση και να καθοριστούν μετρήσιμοι δείχτε που θα επιτρέπουν τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να δοθούν κίνητρα προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να καθιερώσουν κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και εσωτερικούς κανόνες ως προς την απεικόνηση των φύλων. Καταλήγοντας, θα ήθελα να επισημάνω την επίγουσα ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την παροχή ποιοτικών και οικονομικά προσιτών δομών, φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους για την καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον γυναικό στην αγορά εργασίας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ. Thank you so much for your... Ευχαριστώ πολύ για την ε, συμβολή σας. Δανία. Ράσμους με συγχωρείτε, είναι πολύ δύσκολο να μην το... Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργάνωσε αυτή τη συνάντηση. Είναι πολύ σημαντικό να μην μιλάμε μόνο για τα πράγματα, να μην μιλάμε μόνο για δεδομένα και μελέτες. Τα έχουμε αυτά. Ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε ότι υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών και στον κόσμο του πολιτισμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν δράση. Πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχουν ε, δημοσιονομικά στις χώρες μέλη, χρειάζεται να δοθούν περισσότερα για τις γυναίκες. 90% είδαμε των ταινιών πριν από 20 χρόνια γινόντουσαν από άντρε, αλλά και σήμερα ακόμα λίγο πολύ είναι το ίδιο. Πώς θα το αλλάξουμε? Ζητώντας ποσοστώσει. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια αλλαγή, θετικά παραδείγματα, ώστε σε 20 χρόνια από τώρα να μην χρειαζόμαστε πια ποσοστώσει. Να σταματήσουμε τις μελέτες και α περάσουμε στη δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που είπατε. Συμφωνώ μαζί σας, ναι. Νορβηγία τώρα. Τον Την Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη δημοκρατία μας τα μέσα ενημέρωσης και πολλά εξαρτώνται από τους δημοσιογράφους και τις ειδήσει. Είναι πρόβλημα λοιπόν να είναι υπόθεση των ανδρών τα μέσα ενημέρωσης, γιατί και εμείς μπορούμε να έχουμε ένα επικριτικό βλέμμα και αυτιά επίσης σε σχέση με τόσα συμβαίνουν. Άσε που ειδήσει τα νέα δεν έχουν σύνορα. 80% πάντως των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι άντρες σήμερα. Εκεί η διαφορά είναι τεράστια. Και αν αυτό συνεχίζεται, αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί και η ανισορροπία. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί έτσι τα προϊόντα ε, είναι τελικά καταφυνόμενα από τους άντρες, αλλά επίσης λείπουν έτσι και κάποιες δεξιότητες. Η κατανάλωση πολλές φορές αποφασίζεται από αλγόριθμους. Αν τους φτιάχνουν οι άντρες, εννοείται ότι θα υπάρχει στρέβλωση. Τα μέσα ενημέρωσης λοιπόν χρειάζονται περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις για να είναι ανταγωνιστικά στο μέλλον. Αυτό πρέπει να μας κάνει να αποφασίσουμε για περισσότερες γυναίκες. Έπειτα, η παρενόχληση και σε αυτό τον κλάδο είναι το ίδιο σημαντικό όπως είναι και σε άλλους. Υπάρχει εκστρατεία στην Νορβηγία, έγινε έρευνα για την σεξουαλική παρενόχληση στον κόσμο των δημοσιογράφων και φάνηκε ότι οι νέε γυναίκε είναι περισσότερο εκτεθειμένε στην σεξουαλική παρενόχληση. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στα μέσα ενημέρωσης. Για να είναι ένας ασφαλής χώρος να εργάζεται κανείς στα μέσα ενημέρωσης. Η συνδυτοποίηση είναι σαν το γάλα. Κρατάει λίγες μέρες. Μετά τίποτα. Γι' αυτό τέτοιες δράσεις και εκστρατείες πρέπει να ανανεώνονται τακτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρουμανία τώρα. Χριστίνα Γιουριστίτς. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω γαλλικά. Χαιρετίζω πρώτα απ' όλα όλους τους προσκεκλημένους εδώ, όλες τις γυναίκες σήμερα. Εκπροσωπώ τη Ρουμανία. Ναι, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Ευκαιριών ε, στη Ρουμανία, στη Βουλή, τη Ρουμανική. Σήμερα δεν είναι η ημέρα της γυναίκας, είναι η μέρα δικαιωμάτων της γυναίκας. Ο αγώνας της γυναίκας συνεχίζεται για τα δικαιώματά της, για να καλύψει όλα αυτά τα χρόνια διακρίσεων και πόνο που πέρασε. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτά να τα θυμόμαστε μια μέρα το χρόνο, γιατί τις άλλες μέρες δεν το συζητάμε, σήμερα το συζητάμε περισσότερο. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι περισσότερη δράση όλο το χρόνο για να ανακτήσουμε αυτό που έχουμε χάσει εκατοντάδες χρόνια. Μετά θα μεταφέρω το μήνυμά μου στα ρουμανικά για να ακουστεί λίγο και η γλώσσα η ρουμανική σε αυτόν τον διαπολιτισμικό διάλογο που κάνουμε μεταξύ μας. Συνεπώς συνεχίζει η Ρουμανικά η ομιλήτρια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε κάποια σημαντικά δεδομένα. Η Ρουμανία τηρεί τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανισότητας ευκαιριών. Οι γυναίκες συμμετέχουν όλο και περισσότερο στο δημόσιο βίο. Οι μελέτες δείχνουν ότι στις χώρες μέλη οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο και δεν μπορούν να συμμετέχουν εξίσου στον κοινωνικό διάλογο. Είναι και θύματα επίσης ε, κακοποίησης. Έχουμε περάσει πολλά χρόνια κομμουνισμού και σήμερα πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια ψυχολογικά κλισέ για το ρόλο των παραδοσιακών της γυναίκας στην κοινωνία και στην οικογένεια. Έχουμε μια καλή γυναίκα που πρέπει να ασχολείται με την οικογένεια, ενώ ο άντρα είναι αυτό που φέρνει τα χρήματα και παίρνει και τι αποφάσει για την οικογένεια ολόκληρη. Είναι και αυτό ένα κλισέ. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο λοιπόν για την ε, ισότητα που εδρεύει στο Βίλνιους λέει ότι ο αριθμό των γυναικών, των ειδικών που εμφανίζονται στην τηλεόραση είναι πολύ πιο μικρός από τους άντρες. Και αυτό όχι μόνο στη Ρουμανία, αλλά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γυναίκες εκφράζουν την κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι συνήθως οι ειδικοί που θα κληθούν στην τηλεόραση. Γίνονται και συστάσει. Πρέπει να καταπολυθούν τα στερεότυπα γυναικών και αντρών, οι εικόνε πούμε που δείχνουν τι γυναίκε να μαγειρεύουν. Οι γυναίκε καλοντημένε, περιποιημένε κλπ. Επίση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ουδέτερη γλώσσα να μην λέμε κυρία πρόεδρε, να λέμε σκέτο πρόεδρε, να χρησιμοποιούμε ουδέτερο, ουδέτερη ορολογία όσον αφορά τη γλώσσα. Επίσης, όσον αφορά την εργασία της γυναίκας στον κλάδο της τεχνολογίας. Οι πυρογνώμονες σε αυτό το κλάδο, σε υψηλό επίπεδο, έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς. Η κατανομή μεταξύ των δύο φύλων δείχνει ότι είναι 53% άντρες μηχανικοί και 47% γυναίκες. Στη Ρουμανία έχει χρηματοδοτηθεί προσπάθεια μέσω προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτείνει να δουλέψουμε για να υπάρξει καλύτερη παρουσίαση του Πώ είναι οι γυναίκες και αυτό στα μέσα ενημέρωσης. Η αντίληψη δηλαδή για τις γυναίκες να αλλάξει, να μην ακολουθεί τα στερεότυπα και γενικά αλλά και πιο συγκεκριμένα στα μέσα ενημέρωσης. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και κάποιες δράσεις που έχουν αληθεί σε εθνικό επίπεδο για το ρόλο των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Ο, η 8η Μαΐου ορίστηκε η μέρα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η Εθνική Υπηρεσία για την Ισότητα οργανώνει από το 2016 την Εβδομάδα Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που είναι αφιερωμένη στα παιδιά και στους εφήβους, την αγόρια τα κορίτσια. Στις 11 Μαΐου του 2016 Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν σε συζητήσεις σε 11 σχολεία στο Βουκουρεστίου, στο Βουκουρέστι και μίλησαν για την θέση των ανδρών και των γυναικών στη δημόσια προβλήθηκαν ταινίε, οργανώθηκαν συζητήσεις για την ενδοικογενειακή βία, για την παρενόχληση, για τις γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων και έγιναν και διαγωνισμοί για το θέμα της ισότητας. Και αυτό, όπως είπαμε, για μαθητές και φοιτητές. Ένα χρόνο μετά, α, διακόπτη πρόεδρος, δεν έχετε χρόνο. Ε, συνεχίζω μιλήτρια. Στο facebook θα βρείτε επίσης διάφορα. Ολοκληρώνω λοιπόν εδώ και σας εύχομαι καρποφόρες εργασίες και καλά προγράμματα για το μέλλον. Ε, ευχαριστώ και καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν εντάξει, τηρούμε το χρόνο μας, αλλά δεν πρέπει να το ξεπερνάμε. Χρησιμοποιούμε τη τεχνολογία, βλέπετε καλά. Όσον αφορά το slide.doil, το ακροτήριο συμμετέχει στην ε, έρευνα αυτή. Σας ευχαριστούμε όλους. Θα σας πω ποιες είναι οι απαντήσεις για τα, τις δύο πρώτες ερωτήσεις. Στην πρώτη ερώτηση, η απάντηση είναι για το πώς οι γυναίκες έχουν καταγράψει ιστορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο. Το 2017 είναι 35% το 2015. Η, η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση, πιο δημοφιλής, για τους γυναικείους χαρακτήρες στα πιο γνωστά φιλμ της αμερικανικής αγοράς. Με αποκαλυπτική ένδυση ήταν 25,9% η πιο δημοφιλής απάντηση. Δεν τα πήγαμε πολύ καλά στις απαντήσεις. Για τις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις από το σλάιντο. Α, να τη διαβάσω αλλιώς γιατί είναι δύσκολο. Τι νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε για να απεικονίζονται με τρόπο θετικό γυναίκε στα μέσα μαζική ενημέρωση. Αυτή ήταν η πιο δημοφιλή ερώτηση. Κυρία Μπιλγκεχάν, έχετε και πάλι το λόγο. Oui, en fait... Euh, ναι, κοιτάξτε οι εκλογείς, οι τηλεθεατές, άντρες, γυναίκες, έτσι. Πάντα το θέμα είναι θέμα ζήτησης και προσφοράς. Πρέπει να υπάρξει πιο απόλυτη τοποθέτηση των γυναικών, των πολιτών γυναικών που διαβάζουν εφημερίδες, που αγοράζουν εφημερίδες, που παρακολουθούν τα μέσα ενημέρωση στο διαδίκτυο. Οι γυναίκες λοιπόν είναι αυτές που πρέπει να εξηγηθούν, που πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους, όπως λέμε, όπως το μωρό που λέγατε πριν που το ένα κλαίει και απαιτεί να το ταΐσει η μαμά του, ενώ το άλλο περιμένει υπομονητικά. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται σε πολλές χώρες. Ο ίδιος αγώνας είναι. Εγώ όταν είμαι στο Στρασβούργο, εκεί στην συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην Επιτροπή μας για την Ισότητα, Εκεί συμμετέχω εδώ και χρόνια. Είμαι εδώ και 15 χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο και είμαι λιγάκι όπως και εσείς. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, ότι γίνονται κάποια βήματα, αλλά ένα βήμα μπρος, δύο πίσω μερικές φορές. Πραγματικά είναι θλιβερό να βλέπουμε ότι μετά από όσα έχουν κάνει οι γιαγιάδες μας στις χώρες μας, ειλικρινά, ίσως οι γιαγιάδες μας να είχαν κάνει περισσότερα βήματα από ότι τα εγγόνια μας. Όταν βλέπουμε πώς αλλάζει ο τρόπος ζωής, η σκέψη, το μίσος για τον άλλον, πώς ε, έχει εμφανιστεί. Πάντως, ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, να στηρίζουμε τις ιδέες μας και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στις χώρες μας. Χαίρομαι που βλέπω ότι εδώ υπάρχει ισότητα, υπάρχουν πολλές γυναίκες που συμμετέχουν στη σημερινή συνεδρίαση, βέβαια περισσότερες γυναίκες από άντρες, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε όλους τους κλάδους, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στο κινηματογράφο, στις τέχνες, στη μουσική. Αυτό. Μπορούμε. Και πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στις γυναίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Η Μικαέλα τώρα. Τρία λεπτά παρακαλώ, έτσι. Πολύ λίγος ο χρόνος, αλλά σας ευχαριστώ. Και για να κλείσω θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, euh, να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας και να ευχαριστήσω και όλους όσους ε, συμμετείχατε στην ε, συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκυλσούμ Βίγκεχαν για την παρουσίασή της. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν την ίδια άποψη. Θέλουμε να δούμε περισσότερες γυναίκες, περισσότερη γυναικεία παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στη... Στο δικό μου το έργο, στην εκθεσία μου δηλαδή για την ισότητα, των δύο φίλων στα μέσα ενημέρωση, αναφέρω την πεποίθησή μου. Λέω ότι και τα μέσα ενημέρωση αλλά και η κοινωνία γενικότερα χρειάζεται περισσότερο την επιρροή των γυναικών. Βέβαια, τελική έκθεση αποτελεί συμβιβασμό ανάμεσα στι δικέ μου τι ιδέε και τι ιδέε των συναδέρφων μου από τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Κυρία Ροντρίγκε, για παράδειγμα, η οποία συνεισέφερε πολύ στην έκθεση αυτή και την ευχαριστώ πολύ. Οι γυναίκε είναι πιο ευάλωτε και στην εργασία τους λόγω φυσικής ε, διαμόρφωσης. Ε, προτείνουμε λοιπόν στην έκθεση αυτή και λύσεις. Θα σας δώσω λίγα μόνο νούμερα γιατί δεν θέλω να επαναλάβω τέτοια και τέτοια. Πάντως 68% του συνόλου των διπλωματούχων στη δημοσιογραφία είναι γυναίκες. Όμως μόνο 20-30% βρίσκονται στη διαχείριση ή σε διευθυντικέ θέσει στα μέσα ενημέρωση. Δεν είναι ισορροπή αυτό. Οι διαφορέ μισθών μεταξύ αντρών και γυναικών πάντα στα μέσα ενημέρωση είναι 17%. Δεν είναι ισορροπή αυτό. Οι γυναίκες επίσης αναφέρονται πολύ λιγότερο ως ειδικοί, ως εμπειρογνώμονε, ω σχολιαστέ, Πάλι 17% μόνο. Δεν φτάνει. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι οι γυναίκες είναι εξίσου έξυπνες και ικανές όπως και οι άντρες. Έχουν όμως να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολες συνθήκες. Το κύριο πρόβλημα είναι η μικρή ε, αντιπροσώπευση των γυναικών στα μέσα ενημέρωση σε υψηλέ διευθυντικέ θέσει. Κάτι το οποίο επηρεάζει τελικά και το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό των μέσων ενημέρωση και την δομή, την οργάνωση, η οποία δεν ευνοεί τις γυναίκες και τον ε, συνδυασμό της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Στην έκθεσή μας δεν προτείνουμε νέα νομοθεσία, θέλουμε όμως να εκπονήσουμε ή μάλλον να εφαρμόσουμε την νομοθεσία που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας. Την οδηγία δηλαδή κατά των διακρίσεων, την οδηγία για την απασχόληση, την οδηγία για τα οπτικοακουστικά και τα νέα μέσα που έχουμε, την οδηγία ας πούμε για την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματική ε, ζωής που συζητούμε αυτή την εποχή στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν όμως και άλλες δράσεις. Πρέπει να στηρίξουμε, να προωθήσουμε την κατάρτιση για τις επαγγελματίε του κλάδου, να πετύσουμε εσωτερικό κανονισμό Κάποιε από σας το ανέφεραν. Επίσης, να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εκστρατείες όπως εκείνη για το πετή κοσόν σεξίστε που έχει τον τίτλο δηλαδή το ε, σεξιστικό γουρουνάκι. Επίσης να προσπαθήσουμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες το Βέλγιο υπάρχει ένα μητρό ε, ειδικών ε, εμπειρογνωμών, δηλαδή γυναικών, εξπερτάλια λέγεται. Εδώ υπάρχει αυτό στο Βέλγιο. Θα μπορούσε να γίνει και αλλού. Τα μέσα ενημέρωση χρειάζονται λοιπόν περισσότερες γυναίκες και την επιρροή τους. Υπάρχουν πολλές γυναίκες δημοσιογράφοι, πολύ θαραλέες. Και αυτό είναι που θέλω να προσθέσω σε αυτό που ρωτήσατε, πώς μπορούμε να στηρίξουμε τέτοια παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν πολλές πολύ γνωστές γυναίκες και ιδιαίτερα δυνατές. τι είδαμε ανάμεσα στις προσκεκλημένες μας. Θέλω λοιπόν να υποφεληθώ εδώ από την παρουσία της ε, εκπροσώπου του Συμβουλίου από την Τουρκία και εσείς είστε δημοσιογράφος, έτσι. Και όντως υπάρχουν πολλές ε, γυναίκες δημοσιογράφοι στην ε, Τουρκία που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. ή βρίσκονται στη φυλακή. Την απελευθέρωσή τους, τη κυρία Νησάκια παράδειγμα, θέλουμε να ζητήσουμε που καταδικάστηκε στα ισόβια για πολιτικούς λόγους. Ξέρω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη εκεί, αλλά εμεί πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας για να απελευθερωθούν. Χαίρομαι που εδώ μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις, εμπειρίες, να συνομιλήσουμε και ελπίζω το έργο μας να πετύχει. Όπως είπατε κι εσείς, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεννοούμαστε πολύ καλά. Είμαστε 40% γυναίκες και στη διαχείριση συμμετέχουμε εξίσου στις επιτροπές, έχουμε αντιπροέδρους, οι μισές είναι γυναίκες στις διάφορες κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Είναι διαφορετική κατάσταση δηλαδή από αυτή που έχουμε στα εθνικά κοινοβούλια ή στα άλλα θεσμικά όργανα. Ελπίζω λοιπόν στο μέλλον να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνεισφορά σας εδώ και για την συνεργασία σας. Thank you, I was very generous. Σε ευχαριστώ, Μικαέλα. Ήμουν τρομερά γενναιόδορη. Σου δώσα σχεδόν 6 λεπτά. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Μπιλγκεχάν, τη Μικαέλα και όλους σας. Θα αγωνιστούμε για όλες τις γυναίκες που καταπιέζονται στον κόσμο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και χαιρετισμού στις γυναίκες της Αιθιοπίας. Αν κάνετε αυτή την κίνηση θα καταλάβουν. Τώρα, ο λόγος της συντονίστρια του δεύτερου πάνελ, την κυρία Ράγε Madam Commissioner. Κύριε Επίτροπε, αξιότοπα μέλη του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίες και μερικοί κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εγκάρδια στο δεύτερο πάνελ της ειδική ε, συνεδρίας της Επιτροπής μας που θα ασχοληθεί με την ενθάρρυνση των ε, γυναικών και των κοριτσιών μέσω ψηφιακή συμπερίληψη. Καλώ ορίζουμε την κυρία Μαρία Γκάμπριελ, Επιτροπό για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία, που θα μιλήσει. Επίση, ε, την ε, κυρία Ιζασκούμπιλ Μπαου Μπαραντίκα, συνάδελφο από το Άλντε, και θα δούμε και, τη, ή μάλλον που είναι υπεύθυνη για την 62η Σύνοδο του ΟΗΕ και της Επιτροπής του για το καστό των Γυναικών, θα μας παρουσιάσει κάποια σχόλια. Μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν έρθει από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρουν το λόγο και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, κοινωνικοί εταίροι και βεβαίως όλοι οι συμμετέχοντες. Επίσης θα έχουμε και ένα βίντεο μήνυμα από τον κύριο Κάρλος Μέδας, Επιτροπό για την Έρευνα, την Επιστημική και την Κοινοτομία, που θα ανακοινώσει τους τελικούς υποψηφίου για, το για το Ευρωπαϊκό Βραβείο για τις Γυναίκες που Κοινοτομούν. Για να κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα, να κάνω εγώ μια μικρή παρέμβαση στα πολωνικά, οπότε παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας on the second channel. Okay. Thank you very much. Szanowni Państwo, sektor ICT. Κυρίε και κύριοι, ο τομέας της πληροφορικής αναπτύσσεται ταχύτατα και η μισθή είναι πολύ ικανοποιητική. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για τις υπηρεσίες αυτές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι θα, υπάρχουν 200, θα λείπουν 200.000 ειδικοί για τα θέματα πληροφορικής. Οι γυναίκες αποτελούν το 30% των εργαζομένων στον τομέα αυτό και κυρίως με χαμηλούς μισθούς και βρίσκονται στα κατώτερα κλιμάκια της σκάλας. Ε, αν δούμε την κατάσταση πιο προσεκτικά, θα καταλάβουμε ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν λιγότερο τις ε, υπηρεσίες online, τις τραπεζικές, ή χρησιμοποιούν τις, ε, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπορίου λιγότερο, χρησιμοποιούν το ίντερνετ λιγότερο, και σε όλες τις ε, παρουσίες ε, του για το ίντερνετ, το ίντερνετ των πραγμάτων και άλλες εξελίξεις βλέπουμε συνήθως ε, άντρες. Αν εμφανιστεί μια γυναίκα είναι απλώς για να τους φέρει τον καφέ. Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνολογία της πληροφορικής μας δίνουν την δυνατότητα να εισαγάγουμε μεγαλύτερη ευελιξία ευελιξία στην, ε, στο χώρο εργασίας, περισσότερες ευκαιρίε για γυναίκες που θέλουν να καινοτομήσουν, περισσότερες ευκαιρίε για την αντιμετώπιση της, ε, ε, των, ανισοτήτων. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις γυναίκες, την απασχόληση των γυναικών, όχι μόνο στις πλούσιες χώρες και περιφέρειες, αλλά και στις πιο φτωχές περιοχές και στην Ήπεθρο η εκμάθηση νέων ε, δεξιοτήτων, ε, θα, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων θα είναι πραγματικά α, σημαντικό στοιχείο για το μέλλον. Αν υπάρχουν ανισότητες στον τομέα της πληροφορικής που όντως υπάρχουν, αυτό πραγματικά μας κοστίζει κάποια δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο τομέας της πληροφορικής αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για τις γυναίκες και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Απλώς πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιούν τα όργανα που έχουν στη διάθεσή τους. Κάνω λοιπόν έκκληση προς τα κρατημέλη και τις κυβερνήσεις τους να εισαγάγουν ε, υποχρεωτική κατάρτιση πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης από τον υπηαγωγείο. Πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες, πρέπει να έχουν την δυνατότητα να μπορούν να επιλέγουν τη σταδιοδρομία τους στο μέλλον. Και τώρα να σας ε, θυμίσω ότι μπορούμε πάλι να μπούμε στο σλάιντο και να συμμετάσχουμε στα ερωτήματα. Δύο είναι τα ερωτήματα. Ένα είναι ποια μεταξύ των τεσσάρων ε, κρατών μελών θεωρείται ότι έχει τη μεγαλύτερη ε, αναλογία σε γυναίκες στους ειδικού ε, πληροφορικής. Τα τέσσερα κράτη-μέλη είναι Βέλγιο, Εστονία, Σουηδία, Βουλγαρία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο είναι το ποσοστό των, ε, των αποφύτων γυναικών από τα, στον τομέα της πληροφορικής. Τα ποσοστά είναι 9, 17, 29 και 51%. Και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε κάποια ερωτήματα. Αν τώρα όσοι μας παρακολουθούν μέσω του ίντερνετ μπορούν, θέλουν να θέσουν ένα ερώτημα στην ε, ε, Επίτροπο, μπορούν να το γράψουν στο σλάιντο ή μπορούν και να ψηφίσουν για την ε, ερώτηση που προτιμούν και η Επίτροπος θα προσπαθήσει να απαντήσει στο τέλος της, του πάνελ. Οπότε τώρα να καλωσορίσουμε την Επίτροπο Μαρία Γκαμπριέλ. Επίτροπο για την Ψηφιακή Οικονομία και την ε, Κοινωνία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κοσλόφσκα Ράγεβιτς Ανιέσκα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συμμετέχοντες και προσκεκλημένοι, Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε εδώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη Διεθνή ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας. Συγχρόνως έρχομαι εδώ με ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί εδώ και νέα μήνες είμαι Επιτροπός Αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία, αλλά βρίσκομαι εδώ μαζί με ανθρώπους που σας διαβεβαιώ μπορείτε να βασιστείτε σε εμά. Υπάρχουν και ευρωβουλευτές, κάποιοι δεν είναι εδώ, αλλά ξέρω ότι αγωνίζονται για τα δικαιώματα της γυναίκας και τους θαυμάζω για τον τρόπο με τον οποίο στηρίζουν τη γυναίκα και τη θέση της μέσω της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη δύναμη που μας δίνετε γιατί εσείς είσαστε η δύναμή μας. Ποιο είναι το σημερινό μας θέμα λοιπόν να υπενθυμίσω ότι πριν από δέκα χρόνια την Κίνα, την Ινδία, ε, ήταν πράγματα που τα ξεχνάγαμε και η ψηφιακή οικονομία δεν είχε καθόλου μέσα τη γυναίκα. Τα, τις τελευταίες ε, δύο δεκαετίες έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουμε περισσότερη ανάπτυξη στο ΑΕΠ μέσω της ψηφιακής οικονομίας έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο το ΕΠ. Η κοινωνία όμως, από την άλλη μεριά, πρέπει να αναρωτηθεί. Η κοινωνία παίρνει στα σοβαρά αυτό το μέσο ανάπτυξης. Σήμερα ακούμε για τη συνεισφορά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά θα υπογραμμίσω ότι γίνεται στην ε, ψηφιακή οικονομία. Γιατί είμαι υπεύθυνη για αυτό το θέμα βέβαια, αλλά και γιατί με ανησυχεί πάρα πολύ η κατάφορη απουσία των γυναικών σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν αλλαγές στον ψηφιακό κλάδο αποφασιστικής σημασίας. Καλό είναι αυτό, ναι, θετικό και το δείχνουν και τα νούμερα αυτό. Μια ψηφιακή Ευρώπη ε, προσθέτει 15 ε, εκατομμύρια στην οικονομία της, το ΕΠ οι τεχνολογίες εχμής, η ε, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν τις χώρες που είναι περισσότερο ψηφιοποιημένες να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μέχρι το 2020. Για να γίνει αυτό όμως υπάρχει και κάτι που ζητάμε επίμονα. Περισσότερους ειδικού καταρτισμένους στον τομέα αυτής της τεχνολογίας. Μετά το 2020, πάνω από 90% των θέσεων απασχόλησης θα, θα απαιτούν τέτοιες βασικές δεξιότητες στην ψηφιακή τεχνολογία. Τι μπορούν λοιπόν να προσφέρουν σε αυτό το ψηφιακό μέλλον οι γυναίκε. Η απάντηση είναι σαφής. Περισσότερες γυναίκες στην ψηφιακή απασχόληση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση ετήσια του ΕΠ 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να υπάρξει επίσης βελτίωση για το περιβάλλον των startups, γιατί startups ε, που έχουν φτιαχτεί από γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν. Και οι επιχειρήσεις έχουν να κερδίσουν από την ποικιλομορφία. Προσφέρουν καλύτερα προϊόντα και καλύτερες υπηρεσίε. Αυτά είναι τα συμπεράσματα της τελευταίας μελέτης που έγινε για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή που δημοσιεύει σήμερα η Επιτροπή και εγώ είμαι η πρώτη που την αναφέρω και εσείς οι πρώτοι που τη μαθαίνετε. Πολύ σημαντικό λοιπόν για την ανάπτυξη γυναίκε. Πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε ακριβώ. Σε παγκόσμιο επίπεδο η ΕΠ πέρυσι είπε ότι η πρόοδο για την ισότητα βρίσκεται σε νεκρό σημείο και το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων αυξάνεται. Και η μελέτη μα επιβεβαιώνει αυτό το αποτέλεσμα ακριβώ. Τέσσερις φορέ περισσότεροι άντρε από γυναίκε είναι στην Ευρώπη που έχουν καταρτιστεί στα θέματα τεχνολογιών και τα ψηφιακά. Και πιο σημαντικό ακόμα, ο αριθμό των γυναικών στην ανώτατη εκπαίδευση που ασχολείται με την πληροφορική έχει πέσει σε σχέση με το 2011. Και η πτώση αυτή αντικατοπτρίζεται και στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στις σχετικές επιχειρήσεις, του κλάδου δηλαδή, που ακόμα και αν έχουν φτιαχτεί από τις γυναίκες, αυτές τώρα υποχωρούν σιγά σιγά σε θέσεις υψηλά ισταμένων σε κλάδους τεχνολογίας οι άντρες έχουν ε, πέντε φορές περισσότερο την ευκαιρία να βρεθούν σε τέτοιες ηγετικές θέσεις από τις γυναίκες. Και όμως οι γυναίκες είναι όσοι και άντρες στην κοινωνία μας. 19% όμως είναι οι γυναίκες που φτιάχνουν τέτοιες επιχειρήσεις. Ανάμεσα στο 2010 και στο 2015 πολύ λίγες γυναίκες έφτιαξαν τέτοιες επιχειρήσεις. Στην ανάπτυξη επίσης των προϊόντων των ψηφιακών, οι γυναίκες είναι όλο και περισσότερο αποκομμένες από το μέλλον γιατί δεν συμμετέχουν σε αυτά. Αυτό αποτελεί και κοινωνική αδικία αλλά και απώλεια για την οικονομία μας και για την κοινωνία στο σύνολό της. Πώς λοιπόν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα κορίτσια και γυναίκες να συμμετέχουν να αλλάξει η τάση αυτή. Δεν υπάρχει βέβαια κανένα μαγικό ραβδί. Χρειαζόμαστε πολλαπλές λύσεις που να καταπολεμούν τις ρίζες ε, που είναι περίπλοκες. Όλοι καταλαβαίνουμε τι συνέπειες έχουν οι δράσεις μας. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν δράσεις σε κάθε επίπεδο. Οι συνεργάτε μου και εγώ δουλεύουμε πάνω σε μια στρατηγική για την παρουσία των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο που θα βασίζεται σε τρία σκέλη. Πρώτον, να αντιμετωπίσουμε τα παλιά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών που παραμένουν στις κοινωνίες μας και στην ψηφιακή οικονομία. Το γνωρίζουμε όλοι. Η επιλογή της σταδιοδρομίας ε, δεν είναι κάτι γραμμικό σαν απόφαση. Πολλοί παράγοντε επηρεάζουν την απόφαση αυτή. Το κοινωνικό περιβάλλον όπου μεγάλωσε κανεί, η οικογένεια, οι αξίε, οι αντιλήψει και τα μέσα ενημέρωση έχουν λόγο σε αυτό. Γιατί διαμορφώνουν τι πεπιθήσει μα, τι αξίε μα και την αντίληψή μα για την πραγματικότητα. Αν όλες, όλα τα κορίτσια ακούσουν στα μέσα ενημέρωση ότι οι τεχνολογίε πληροφοριών και οι επικοινωνίε είναι για τα γόρια, που τους αρέσει να απομονώνονται και να δουλεύουν σε αυτά, ενώ δεν είναι κάτι θηλυκό, ε, δεν θα το διαλέξουν. Οι γυναίκες, οι άντρες, τα γόρια δεν, ε, ε, και τα κορίτσια δεν εκτίθενται πάντα στην πραγματικότητα. Όταν λοιπόν δεν βλέπουν οι γυναίκες σε αυτό τον κλάδο, δεν τον ακολουθούν. Στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι 80% γυναίκες, 26% στα tweet και στο διαδίκτυο. Επιπλέον, δεν βλέπουν ε, γυναίκες που εμφανίζονται με θετική εικόνα. Η σταδιοδρομία ε, που ανθίζει για γυναίκες είναι πολύ λίγες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν εδώ τίθεται θέμα προβολή των γυναικών. Σε μελέτη της Microsoft φάνηκε ότι οι γυναίκες δεν θέλουν να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες επιστημών, μαθηματικών, τεχνολογίας κτλ. παρόλο που γνωρίζουν τα θετικά για να βρουν δουλειά στη συνέχεια. Και η μελέτη μας επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες όντως ε, απέχουν από τέτοιες σταδιοδρομίες γιατί ακριβώς δεν έχουν αντίστοιχα πρότυπα στη ζωή τους στις ταινίε, στη τηλεόραση, στα κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει να παρουσιάζεται σωστά η εικόνα της γυναίκας και ο ρόλος που μπορεί να παίξει στην κοινωνία. Οι χώρες μέλη λοιπόν έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν από αυτού. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Η οδηγία για το οπτικοακουστικά. Διαπραγματευόμαστε τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ε, στην τη της οδηγίας αυτής, όπου απαγορεύεται η διάκριση εξαιτία του φύλου στις ε, εμπορικές διαφημίσεις. Το 2016 υπήρξε σύσταση επίσης για την προστασία των ανηλίκων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και όλα αυτά σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων Ζητάμε από τις επιχειρήσεις να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και να παρουσιάσουν μια εικόνα διαφοροποιημένη και ρεαλιστική όσον αφορά τις δυνατότητες και τις ικανότητες των ανδρών και των γυναικών στις κοινωνίες μας. Θέλω να δω τι κάνουν οι χώρες μέλη σε αυτά και να συζητήσω μαζί τους για τα αποτελέσματα και με τους εθνικούς ρυθμιστές και τους κλάδους. Η υποεκπροσώπηση πάντως των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης μας εκπλήσει τελικά, δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς στον κλάδο των οπτικοακουστικών υποεκπροσωπούνται. Αν οι ταινίε, ε, τα βιντεοπαιχνίδια, ε, οι διάφορες εκπομπές προετοιμάζονται από τις γυναίκες, πώς να έχουμε μια πιο διαφοροποιημένη εικόνα. Χρειάζεται περισσότερη ισορροπία λοιπόν μεταξύ των δύο φύλων στα οπτικοακουστικά, στα μέσα ενημέρωσης, να δώσουμε περισσότερο χρώμα και διαφοροποίηση στην πολιτιστική μας παραγωγή. Ίσως κάποιοι να πιστεύουν ότι είναι λογικό οι άντρες και οι γυναίκες να παίζουν ρόλο στα οπτικοακουστικά. Ναι, αλλά όταν ε, το πιστέψει αυτό κανείς, τότε θα διαλέγει ανάλογα και τις σπουδέ που θα ακολουθήσει, για να το πω απλά. Αν δείτε το μοντέλο, το πρότυπο, θα κατευθυνθείτε και προς αυτή την κατεύθυνση. Δουλεύουμε λοιπόν για τέτοια προγράμματα και ευχαριστούμε πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξή του. Από την αρχή έχουμε το πρόγραμμα Media, που είναι μια πραγματική επιτυχία για μας τα καταφέραμε και γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το προωθεί και το στηρίζει και θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να έχουμε χρήματα και στον επόμενο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δουλεύοντας πάντως πάνω σε αυτό το πρόγραμμα ε, Media, θα αναλύσουμε ποια είναι η εκπροσώπηση τελικά των γενικών στα διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούμε. Αυτό κάνουμε αυτή την εποχή, γιατί προσπαθούμε να δούμε μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει στο πρόγραμμα Media για την επόμενη περίοδο 2018-2020. Θα οργανώσουμε επίσης και, και μια εκδήλωση στο Φεστιβάλ των Κανών το 2018, συνεργασία με διάφορου εταίρους, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σε αυτό το ζήτημα. Προβλέπω και άλλε δράσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έτου πολιτιστική κληρονομία και του Ευρωπαϊκού για παράδειγμα, θα είναι κομμάτι της στρατηγικής που θα παρουσιάσω σύντομα. Στα πλαίσια του Ρεπάνα, γιατί να μην θυμηθούμε τι έγινε όλες αυτές τις δεκαετίες και πώς ενισχύθηκαν τα δικαιώματα της γυναίκας. Να βοηθήσουμε φόρο τιμής στις γυναίκες αυτές που πάλεψαν για να δείξουμε ότι η γυναίκα δεν είναι θύμα, είναι αυτή που παίρνει το μέλλον της στα χέρια της. Το καταλάβατε, το βασικό είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε όλα τα επίπεδα. Για μένα, έτσι κι αλλιώς είναι η μόνη επιλογή για να αλλάξουν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Πρέπει να δυναμώσουμε τη φωνή μας, να παρουσιάσουμε περισσότερα γυναικεία πρότυπα. Τα μέσα ενημέρωση αναφέρονται στο τύπο ένας και άλλος πυρογνώμων άντρας. Όχι, πρέπει να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες στα διάφορα πάνελ. Εδώ βέβαια εντάξει έχουμε περισσότερες γυναίκες στα σημερινά πάνελ. Είναι μια εξαίρεση. Το 2018 δεν πρέπει να δεχόμαστε πια πάνελ που να έχουν μόνο άντρε. Πρέπει να συμμετέχουν και γυναίκες. Εξού και τη Δευτέρα που μας πέρασε ξεκίνησα μια εκστρατεία που λέγεται No Women, No Panel και δεσμεύτηκα να μην συμμετέχω σε διασκέψεις και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις όπου δεν υπάρχουν και γυναίκες στα αντίστοιχα ε, πάνελ. Ή όπου θα είμαι η μόνη γυναίκα, δεν το θέλω αυτό. Λοιπόν, σας παρακαλώ να μας στηρίξετε κι εσείς αυτή την εκστρατεία και να διαδώσετε αυτό το μήνυμα. Στην καρδιά του προβλήματος, ξέρουμε τη βρίσκεται. Πάντως ένα από τα συμπεράσματα τη μελέτη μας είναι ότι συχνά ο αποκλεισμό των γυναικών δεν γίνεται επίτηδε. Είναι υποσυνείδητα που γίνεται. Οι γυναίκε έτσι κι αλλιώ είναι απούσε σε πολλέ διασκέψει τόσα πολλά χρόνια που οι οργανωτέ δεν σκέφτονται καν να καλέσουν γυναίκε. Είμαστε αποφασισμένε λοιπόν να αποτελέσουμε το παράδειγμα και να στηρίξουμε το αν δεν υπάρχουν γυναίκες δεν θα υπάρχει ούτε και πάνελ. Η διάκριση δεν έχει θέση εδώ ούτε βέβαια και οι ποσοστώσει, αλλά θέλουμε να οργανώνονται εκδηλώσει που να αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν αρκετές ικανές γυναίκες για να εμφανιστούν στα πάνελ τους. Η μόρφωση εδώ είναι βέβαια βασικό στοιχείο. Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να φροντίσουμε για τέτοια παραδείγματα. Την πρόκληση αυτή όμως πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και έτσι ώστε το ψηφιακό στοιχείο να δώσει περισσότερη δύναμη στις γυναίκες. Για την μόρφωση που έλεγα πριν, 90% των κοριτσιών ενδιαφέρονται για τις τεχνολογίες πληροφορικής. Παρ' όλα αυτά, δεν θα ακολουθήσουν τέτοιες σπουδέ στο πανεπιστήμιο, παρά το ενδιαφέρον αυτό που δείχνουν. Σήμερα λοιπόν η έκθεση μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να αλλάξουν, να συμμετάσχουν περισσότερο σε σαδιοδρομίες σε πληροφορικής, ώστε να αναλάβουν και πρωταγωνιστικό ρόλο αργότερα όταν ε, αποκτήσουν ένα επάγγελμα. Πάντως, το καλό είναι ότι με πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε τον Επίτροπο των Ομόδων για την εκπαίδευση, τον Ιανουάριο παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα δράσης για την μόρφωση στην πληροφορική. Σήμερα θέλουμε να ενθαρρύνουμε να γίνει καλύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ώστε τα κορίτσια, οι γυναίκες, να αποκτήσουν τις κατάλληλες και αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες. Υπογραμμίζουμε ότι τα νέα κορίτσια στην Ευρώπη πρέπει να μάθουν τους βασικούς αλγόριθμους, πρέπει να αποκτήσουν τις βάσεις για να μπορέσουν να δημιουργήσουν στο μέλλον. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η νέα μου φιλοδοξία είναι η εβδομάδα του κώδικα. Κάθε Οκτώβριο δηλαδή, όλο τον Οκτώβριο, κάθε χρόνο, να έχουμε πρωτοβουλία με θελοντές, ώστε να μαθαίνουμε όχι μόνο στους νέους τι είναι κωδικοποίηση. Να τους εξηγήσουμε ότι δεν είμαστε μόνο χρήστες περιεχομένου, αλλά είμαστε και δημιουργοί. Τα μηχανήματα δεν θα αντικαταστήσουν ποτέ πλήρως τον άνθρωπο στην δημιουργία. Γι' αυτό και χαίρομαι όταν βλέπουμε τα νούμερα. Κάθε χρόνο διαπιστώνουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερο συμμετέχοντες, 1,2 εκατομμύρια είχαμε φέτος και 40% ήταν Μεγάλο το ποσοστό. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια. Είχα την ευκαιρία να το πω, αλλά το μοιράζομαι και μαζί σας. Φιλοδοξία μου είναι να έχω 50% των σχολείων στην Ευρώπη ε, μέχρι το 2020 που να συμμετέχουν στην εβδομάδα αυτή του κώδικα. Να ξέρετε ότι θα στηριχτώ στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις ε, δεξιότητες στον ψηφιακό κόσμο βασιζόμαστε σε 19 εθνικές συμμαχίες. Όσες χώρες δεν συμμετέχουν, παρακαλώ να το σκεφτούν και να συμμετάσχουν. Σε ένα χρόνο η συμμαχία αυτή πρόσφερε σε 7 εκατομμύρια Ευρωπαίους κατάρτιση στην ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό δείχνει ότι χρειάζεται κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα δεν θα είναι μόνο οι χώρε μέλη, δεν θα είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κοινωνία των Πολιτών. Όχι, πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι υπέρ των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτή είναι η βαθιά μου πεποίθηση. Και γι' αυτό και αποτελεί προτεραιότητά μου, είναι η προτεραιότητα αριθμός 1 για μένα. Αν προτείνουμε τα καλύτερα νομοθετικά κείμενα, αν έχουμε τα κατάλληλα κονδύλια αλλά αν δεν επενδύσουμε στους άντρες και στις γυναίκες σήμερα, αυτή η ψηφιακή μετάβαση δεν θα οδηγήσει ποτέ στα θετικά αποτελέσματα που όλοι θέλουμε. Έχουμε και άλλα. Ο Επίτροπος Μοέδας μας μίλησε για το βραβείο της καινοτομίας. Τα βραβεία που αποδίδονται σε πρωτοβουλίες των ειδικών ε, των ε, τεχνολογιών πληροφορικής ή πέρσι το IT4C ή τέλο πάντων για την πρόθεση των ψηφιακών δεξιοτήτων ε, κοριτσιών και γυναικών. Θα καλέσω τα κράτη-μέλη να δράσουν σε εθνικό επίπεδο και πραγματικά ελπίζω ότι μπορούμε να υπολογίσουμε σε αυτό. Τρίτη προτεραιότητα, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα και η καινοτομία η έλλειψη κρίσιμης μάζας κοριτσιών και γυναικών στην εκπαίδευση ε, του κλάδου αυτού έχει οδηγήσει σε έλλειψη επαγγελματικών σταδιοδρομιών στον τομέα των ICT. Είναι δύσκολο επίσης όταν ξεκινήσει μια γυναίκα τέτοια καριέρα να μείνει και να προοδεύσει. 17% μόνο των γυναικών που εργάζονται, ε, των απασχολούμενων στον τομέα αυτό είναι γυναίκες. Ταυτόχρονα η Ευρώπη έχει έλλειψη ειδικότητα ε, σε ITC. 40% των επιχειρήσεων που ψάχνουν ε, εμπειρογνώμονε ε, στον τομέα αυτό λένε ότι έχουν τεράστια δυσκολία για να προσλάβουν αυτούς που χρειάζονται. Ένα παράδειγμα που ευνηδιάζει. Ο τομέα τη κυβερνοασφάλεια είναι ένα παράδειγμα όπου υπάρχει σοβαρή έλλειψη γυναικών με ε, ικανότητες και προσόντα και η έλλειψη αυτή φτάνει το 1,8 δις ε, θέσεις απασχόλησης μέχρι το 2022 και 350.000 θέσεις θα βρισκόνται μόνο στην Ευρώπη. Μπορώ λοιπόν να σας βεβαιώσω ότι αυτήν ε, την έλλειψη δεν την καλύψουμε μόνο με άντρες. Επίσης, σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες και στον κλάδο αυτό. Θα πρέπει και πάλι να αναρωτηθούμε τι εμποδίζει τις γυναίκες να δημιουργήσουν εταιρείε τεχνολογίας ή να αρχίσουν να ασχολούνται με τη διαχείρισή τους. Υπάρχει έλλειψη προτύπων για να αισθανθούν αυτοπεποίθηση. Για να, ε, η έλλειψη αυτοπεποίθησης επίσης είναι πάντοτε κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, εδώ πρέπει και το δίκτυο των επιχειρήσεων να στηρίξει τις γυναίκες. Χρειάζεται και κάποια οικονομική στήριξη που μέχρι τώρα είναι αδύναμη. Σύμφωνα με, την, ε, τον Οργανισμό για τις Επιχειρήσεις της Ευρώπης, μέχρι τώρα μόνο 6% των ε, επιχειρήσεων στην Ευρώπη στον τομέα IB έχουν γενικούς διευθυντές γυναίκες. Οι οικονομικές μελέτες δείχνουν ότι οι επενδύσεις στις νεοφυείς επιχειρήσεις ε, από, που έχουν ιδρυθεί από γυναίκες έχουν 63% καλύτερα αποτελέσματα από τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει άντρε. Στον τομέα της συνεργατικής χρηματοδότησης, οι εκστρατείε που έχουν ξεκινήσει οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία από τις εκστρατείες που ξεκινάνε οι άντρε. Με 10 και 13% ποσοστά επιτυχίες συνολικά. Η δράση των γυναικών στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα είναι για μα προτεραιότητα. Παρ' όλα αυτά δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρηματοδότησε 8 hub. Την πρώτη ευρωπαϊκή κοινότητα για την διασύνδεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ώστε να υποστηριχθούν οι γυναίκες επιχειρηματίες στον ε, ψηφιακό κλάδο. Επίσης το βραβείο ε, για τις ε, καινοτόμες γυναίκες βραβεύει τις γυναίκες που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και τις κάνει πρότυπα για τις υπόλοιπες. Ε, εδώ ο στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε και τον, την κοινότητα των ερευνητών ε, και της όλης κοινότητας των ε, όσων εργάζονται στον τομέα ICT. Το ίδιο και στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Εκεί θέλουμε να πετύχουμε κάποια ισορροπία. Θέλουμε να βοηθήσουμε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται. Όταν μιλάμε για κυβερνοασφάλεια, η έλλειψη δεξιοτήτων για τις γυναίκες σημαίνει κίνδυνο για την ασφάλειά μας, για την οικονομία, τη δημοκρατία, για τις κοινωνίες μας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις τρέχουσες πρωτοβουλίες, ώστε ταυτόχρονα να ε, εργαστούμε για να καταπολεμήσουμε τις αρνητικές προκαταλήψεις από τις οποίες υποφέρουν οι γυναίκες από τον τομέα, αλλά και να τις υποστηρίξουμε. Φυσικά ο διάλογος με τις επιχειρήσεις, με τα κάτι μέλη, με τις κοινότητες των ερευνητών, είναι ε, ένα μέσο που πρέπει να αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε πιστικά αποτελέσματα. Και τέλος, το τελευταίο, να μην ξεχνάμε τη διεθνή διάσταση. Το Κοινοβούλιο ποτέ δεν την χάνει αυτήν την προοπτική και είναι οι αξίες και οι αρχές μας αυτό που προασπιζόμαστε όπως ή άλλως, δεν έχουμε επιλογή. Όμως να μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες δεν είναι ένα ομοιογενές ε, μερίδιο του πληθυσμού, όπως δεν είναι και οι χώρες. Πρέπει να ε, βλέπουμε τις γυναίκες και εντός της Ένωσης αλλά και εκτός. Στα πλαίσια της ψηφιακής πολιτικής για την ανάπτυξη λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε τους εταίρους μας να στήσουν περισσότερα προγράμματα τα οποία μπορεί να δώσουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να έχουν απασχόληση και μια σχετική προοπτική. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Ανάπτυξη τον Ιούνιο θα συμπεριλάβει ένα πάνελ ε, με θέμα τη γυναίκες και τα κορίτσια στον χώρο τη ψηφιοποίηση, διότι εκεί θέλουμε να δώσουμε έμπνευση και κίνητρο στι γυναίκε και τα κορίτσια. Για να ολοκληρώσω, στη σημερινή ημέρα της 8 ε, Μαρτίου για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων, έχω ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Χρειαζόμαστε την δέσμευση ανδρών, γυναικών, σχολείων, πανεπιστημίων, εταιριών, του Ευρωκοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, των κρατών μελών, για να πετύχουμε τους στόχους μας. Το Ευρωκοινοβούλιο ανέκαθεν ναι, έκανε πολλά στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Όπως καταλάβατε, είναι ένα θέμα που μου είναι εξαιρετικά προσφυλές. Ε, ήμουν ιδιαίτερα μακροσκελής, αλλά μιλάω από καρδιάς και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς και θα πρέπει να πω από καρδιάς και πάλι ότι δηλώσεις μας και τα λόγια πρέπει να συνοδεύονται από πράξεις. Η αξιοπιστία μας είναι αυτό που, διακυβε... αντικείμενο, αυτό που εδώ διακυβεύεται. Εδώ λοιπόν ε, σας στέλνω την απαραίτητη ενέργεια και ελπίζω να δείξουμε όλοι ε, τον δυναμισμό που χρειάζεται, ώστε η εκφράσεις που και τα λόγια μας σήμερα να ε, μεταφραστούν σε πραγματικότητα. Θέλω να γίνουν πράξη όσα είπαμε. Και πραγματικά ε, θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ έναν κόσμο που η ψηφιακή επανάσταση θα διαφυλάξει παρόλα αυτά το πλέον σημαντικό το ανθρώπινο «ον» και το ανθρώπινο πρόσωπό της. Αυτό το πρόσωπο κατ' εμέ, το ενσαρκώνουν τόσο οι άντρε όσο και οι γυναίκε. Να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Madam Commissioner, for... Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Επίτροπε. Μας ενέπνευσαν τα λόγια σας. Τώρα θα δούμε το βίντεο μήνυμα του Επιτρόπου Μέδας για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και εύχομαι ότι καλύτερο για την Διεθνή ημέρα της γυναίκας. Η επιτυχία σας δεν θα καθοριστεί από το φίλο σας, αλλά μόνο από το πόσο ευρεία είναι το όνειρά σας και πόσο σκληρά θα δουλέψετε για να τα πετύχετε. Αυτά είναι τα λόγια της πιο διάσημης αρχιτέκτονος, της Ζάχα Χαντίντ, πριν πεθάνει. Ε, τη μέρα αυτή λοιπόν ο κόσμος ε, φωνάζει το πόσο σημαντική είναι η ισότητα των φίλων. Πολλοί από εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, αυτό το κάνετε τη δική σας αποστολή για κάθε μέρα του χρόνου. Για μένα η μάχη αυτή πρέπει να κερδιθεί σε πολλά μέτωπα. Και δύο από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας είναι η επιστήμη και η κοινοτομία για να τα καταφέρουμε. Και αυτό είναι το πραγματικό πνεύμα του Ευρωπαϊκού Βραβείου για τις γυναίκες που κοινοτομούν. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να καταδείξουμε όλες τις πτυχές και όλες τις γυναίκες στην κοινοτομία. Φέτος λάβαμε 122 αιτήσει. Κάθε μία ήρθε από μια πραγματικά εξαιρετική γυναίκα ε, σχετικά με τις καινοτομίε της. 26 Ιουνίου στην ε, διάσκεψη Webbit στη Σόφια θα ανακοινώσω τους νικητές. Και σήμερα εδώ μπροστά σας μπορώ να σας ανακοινώσω τις 12 τελικούς ε, υποψηφίους. Πριν όμως το κάνω πρέπει να πω ευχαριστώ στην Επιτροπή Γυναικών και κυρίως στην Πρόεδρό σας, την Βιλίτσια Μπλίνκεβιτσιούτε η, αποστολή σας και η επιμονή σας για να επιτύχετε είναι πραγματικά άξια επένου. Δεν θα σας κρατήσω άλλο, κυρίες και κύριοι, σας που ήρθατε σήμερα από τις τέσσερις ε, γωνιές της Ευρώπης. Βλέπετε τώρα τις 12 τελικές υποψηφίους για το βραβείο καινοτομίας για το 2018. I'd like to uh, Συγχαρητήρια λοιπόν στις 12 ε, τελικές υποψηφίους για, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Βραβείο. Τώρα, μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θα δώσω το πολύ δύο λεπτά στον καθένα που θέλει να μιλήσει και έχω και σφυράκι και θα το χρησιμοποιήσω εάν χρειαστεί. Λοιπόν, ξεκινούμε από την Ισπανία. Σουζάνα Καμέρο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τι εισηγήτριες για την ανάγκη παρουσίας των γυναικών ε, στον ψηφιακό κόσμο. Ε, ρωτούσε και ο Επίτροπο τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω εμείς στην Ισπανία τι κάνουμε. Από το 2014 έχουμε πρόγραμμα δράσης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον ψηφιακό κόσμο και στην κόσμο της πληροφορίας. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να το πετύχουμε αυτό και συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες και οργανώσεις για να δώσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις γυναίκες, στις νέες τεχνολογίες και προκειμένου να αντιμετωπιστούν ματσιστικές συμπεριφορές και παρενόχληση εκεί. Στην εργασία, όπως λέτε, προτείνεται περισσότερη συμμετοχή των γυναικών στις τεχνολογικές θέσεις απασχόλησης και στις διευθυντικές. Στην Ισπανία, να ξέρετε, ότι οι γυναίκες είναι επικεφαλής στην Google, την Microsoft, στο Twitter, Facebook. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Η μόρφωση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όντως, δεν εκπροσωπούνται αρκετά στον πιο κόσμο γυναίκες παρόλο που είναι το μέλλον. Πρέπει επίση να αντιμετωπίσουμε ματζεστικές συμπεριφορέ στο περιεχόμενο, στα βιντεοπαιχνίδια, όπου παραμένουν ε, τα στερότυπα των ρόλων των δύο φύλων. Και επίση και στην ύπεθρο να φροντίσουμε να εξοπλίσουμε τι γυναίκε με ε, νέες δυνατότητες ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία είναι σημαντικό και για το επαγγελματικό τους μέλλον, αλλά για να αποφύγουν και την απομόνωση επίσης για να αντιμετωπίσουν και την ενδοοικογενειακή βία. Θέλω να σας πω ότι στην Ισπανία ε, μόλις υπογράψαμε ένα ιστορική σημασία σύμφωνο για την καταπολέμηση των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων που απευθύνεται κυρίως στους νέους μας, γιατί αυτοί μας απασχολούν πιο πολύ, γιατί εκεί παραμένουν μερικές φορές ε, ματσιστικές συμπεριφορές. Η εκπαίδευση των νέων, Επίσης η κατάρτιση των ε, διδασκόντων έχει μεγάλη σημασία ώστε αυτοί που θα γίνουν ε, πατεράδες να συμπεριφερθούν καλύτερα από εδώ και πέρα. Έχουμε και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να μάθουμε στις νέες και στους νέους μας να αναγνωρίζουν ε, συμπεριφορές ματσιστικές ε, να μάθουν να τις σταματάνε, να τις αποφεύγουν και να πάψει έτσι ο φαύλος κύκλος του, της ματσιστικής συμπεριφοράς. Επίσης φροντίζουμε νομοθετικά να περάσουμε τους νόμους που χρειάζεται για να πάψει αυτή η ψηφιακή βία. Όπως είπαμε, προσβολές ε, και τα λοιπά στον ψηφιακό κόσμο, στο διαδίκτυο, και επίσης ε, να υπάρχουν και κυρώσεις και τιμωρία. Λοιπόν, όσο περισσότερες γυναίκες είναι στον ψηφιακό κόσμο, τόσο περισσότερη δημοκρατία θα έχουμε τελικά στις χώρες μας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Καμαρέρο. Από την Τσεχία τώρα. Φραντίστακ Κοπρίβα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σόιντροβα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δουλειά που έχουν κάνει. Δεν ξέρω αν είμαι ειδικό στον τομέα αυτό, αλλά ήρθα σε επαφή με τους συναδέλφους μου και συμφωνώ σε σχέση με τα όσα είπανε για το περιεχόμενο της έκθεσης. Όντως, πρέπει να καταρρύψουμε τα εμπόδια. Πρέπει να πω ότι οι ποσοστώσεις δεν θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος για να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί οι ποσοστώσεις μπορούν να, επι... να υποχρεώσουν τις γυναίκες να μπουν σε μια θέση που δεν αισθάνονται άνετα. Για παράδειγμα, μια γυναίκα που έχει πάρει μια θέση λόγω ποσόστοσης, μπορεί να θεωρεί ότι οι άλλοι τη θεωρούν ακριβώς ότι έχει τη θέση αυτή λόγω της ποσότητας που πήρε και όχι επειδή είναι ικανή να την κατέχει. Θεωρώ ότι ο δημόσιος τομέας πάντα πρέπει να λαμβάνει τον ηγετικό ρόλο. Και θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα που θα βοηθήσουν τις γυναίκες ας πούμε, να είναι εύκολο για αυτές να φέρουν τα παιδιά τους ή τα μωρά τους, αν έχουν, στη, στο χώρο εργασίας τους. Αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμο από το να πάρουν μια θέση με ποσόστοση. Είναι γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι αρκετά πατριαρχικός και νομίζω ότι πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή ακριβώς στους κλάδους αυτούς όπου γίνονται θετικά πράγματα. Και επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε και όσες έχουν βοηθήσει για να είμαστε τόσο μπροστά στον χώρο της ε, ε, πληροφορικής. Και βεβαίως πρέπει οι γυναίκες να πληρώνονται πολύ καλύτερα και να την χάνουν καλύτερης μεταχείρισης. Να ακούσουμε τώρα την κυρία Γκόμες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Επίτροπε. Είναι μεγάλη μας χαρά να σε έχουμε μαζί μας και που μπορέσαμε να απολαύσουμε την ομιλία σου. την αποφασιστικότητά σου και την έκκληση να μην συμμετέχουμε σε συνεδριάσεις και διασκέψεις χωρίς ίση ε, εκπροσώπηση γυναικών, δηλαδή όχι μία και μόνη προσκεκλημένη. Ε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Χρειαζόμαστε μια και μονη υποστηκλημενη ε ηθελα να ρωτησω το εξης χρειαζομαστε Μια φωνή της Ευρώπης. Μια φωνή που θα ε, προωθήσει την ισότητα των φύλων, θα καταδικάσει κάθε μορφή ανισότητας, διοικητικής μεταχείρισης και παραβίασης γυναικών ε, δικαιωμάτων που είναι εις βάρος των γυναικών στην Ευρώπη και οπουδήποτε στον κόσμο. Πρέπει να πω ότι στην Euronews ε, βλέπουμε ότι πολλές φορές πολλοί το αντιλαμβάνονται αυτό στη φωνή της Ευρώπης όμως στις ειδήσει, ας πούμε, στο του Today, ακριβώς ε, στη σημερινή εκπομπή για την ε, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Άκουσα μια είδηση για τις γυναίκες και καλά ότι στη Σαουδική Αραβία οδηγούν. Εγώ πήγα πρόσφατα και αυτό δεν συνέβαινε καθόλου. Η κυδαιμονία είναι ήδη ε, μια προσβολή στις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας και όχι μόνο, γιατί δεν είναι κάτι που μένει στα χαρτιά. Και είδα, λέει, μια εταιρική σχέση και την Μπάρμπι να ε, προωθείται ως σύμβολο του Σύρος και όχι του Heroes anymore ε, πια για να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού, CNH στη λέξη αυτή. Γιατί η θέση των γυναικών λοιπόν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Μαρία, ήθελα να δώσεις ε, ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το εργαλείο που δεν μπορούν, θα να χρησιμοποιήσουμε μόνο για αυτόν τον σκοπό, ε, για την διάδοση ψευδών ειδήσεων, για τα εργαλεία πληροφορικής, ε, όλα αυτά τα εργαλεία που χρηματοδοτούμε, Καλό θα ήταν να σέβονται την ε, ελευθερία της δημοσιογραφίας και να προωθούν τις ίδιες αξίες με σένα και τις οποίες, στις οποίες προσυπογράφω πλήρως. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Και τώρα από την Πορτογαλία, η κυρία Εστρέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο που θέλω είναι να ε, ευχαριστήσω την Επιτροπή των Γυναικών για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης και να θυμίσω ότι και εγώ ε, ήμουν πρόεδρος εδώ επί 10 χρόνια και είχα τη χαρά να ψηφίσουμε μια σειρά από εκθέσεις. Μπόρεσα σήμερα να ξανασυναντήσω συναδέλφους, συντρόφους από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, όπως τη Μαρία Γκάμπριελ, όπως την κυρία Μπιλμπάο Μπαραντίκα ή την κυρία Μπλινκεβιτσιούτε. Ε, Πράγματι, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Χρειάζονται περισσότερες γυναίκες της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και της πληροφορικής. Χρειάζονται περισσότερες γυναίκες στην ψηφιακή οικονομία. Αυτό ήδη υπόθηκε, αλλά θέλω να το τονίσω. Οι γυναίκες ε, ε, προσωπούνται λοιπόν αυτούς τους κλάδους, ιδιαίτερος σε ό,τι αφορά στις θέσεις ευθύνης. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το 9% δεν αρκεί αυτή η εκπροσώπηση. Στη χώρα μου, στην Πορτογαλία, η είναι το 54%. Όμως στις σχολές ICT είναι μόλις 18%. Και το είπε και η Επίτροπος. Ε, οι νέοι δεν εκδηλώνουν ιδιαίτερη διάθεση να σπουδάσουν σε αυτού του κλάδου. Στην Πορτογαλία όμω είχαμε πολλέ γυναίκε, ευτυχώ, πολλέ γυναίκε επιχειρηματίε, οι οποίε ε, ενεργοποιούνται και στην ψηφιακή οικονομία και στι νεοφυεί επιχειρήσει. Και η Πορτογαλία έχει επενδύσει ιδιαίτερω ε, στην ψηφιακή κοινωνία και την επιχειρηματικότητα εκεί και την ενδυνάμωση, τη χειραφέτηση των γυναικών με μέτρα στήριξη για τι γυναίκε επιχειρηματίε. Εκπαίδευση, καινοτομία, ε, ε, επιστήμε είναι πολιτικέ προτεραιότητε ε, του Πορτογαλικού κράτου. Από πολύ καιρό η τεχνολογία έχει μετατρέψει τις ζωές μας και αυτό συνεχίζεται με γοργό ρυθμό. Η λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση ε, ε σηματοδοτεί βήματα προόδου σε τομείς όπως η ρομποτική και η τεχνητή ευθεία, αλλά οι αλλαγές αυτές ε, έχουν και επιπτώσεις τις οποίες δεν προλαμβάνουμε πάντοτε, όπως με την απασχόληση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη συνδυασμένη αντικτύπο αυτών των ε, φαινομένων. Θα πρέπει να δούμε, θα υπάρξει μαζική καταστροφή θέσεων εργασίας, ένα και περισσότερων, ιδίω θέσεων εργασία για τις γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο απαραίτητο είναι να προβλέψουμε μέτρα για να αποφύγουμε να χάσουμε θέσεις εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, και να μην τις συμπληρώσουμε με αυτά που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο ψηφιακής επανάστασης. Επίσης να πω ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν και πολλές ε, δυνατότητες άσκησης βίας και εκφοβισμού κατά των γυναικών. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη και να το αντιμετωπίσουμε με τα μέτρα που διαθέτουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Στρέλα. Και τώρα από την Πολωνία η κυρία Μπαρόβιτς. Ε, Αγκάτα, przepraszam. Sorry. Ε, Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. E- Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω μιλώντας για κάποιες πολύ χρήσιμες πρωτοβουλίες που έχουμε στην Πολωνία για τα κορίτσια στην εκπαίδευση, για τα κορίτσια που σπουδάζουν επιστήμες πληροφορικής. Έχουν υπάρξει πολλές εκστρατείες ευαισθητοποίηση τέτοιου είδου, έτσι ώστε να υπάρξει, να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην πληροφορική και γενικότερα στι επιστήμε. Έχει υπάρξει μια αύξηση από το 30% στο 37% τα τελευταία χρόνια στον αριθμό των κοριτσιών που εγγράφονται σε τεχνικά, τεχνολογικά πανεπιστήμια. IT for She είναι ένα project που κέρδισε και ένα διαγωνισμό για την κατηγορία ψηφιακές εφαρμογές για γυναίκες. Και μάλιστα η Επίτροπος Γκάμπριελ ε, έδωσε το αντίστοιχο βραβείο. Αυτό το project είναι πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη υπόθεση και μάλιστα ε, αυτή τη χρονιά, το Νοέμβριο, θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση για την παρουσίαση του ρόλου των γυναικών στις, ε, στην τεχνολογία. Ε, θα είναι η Σύνοδος Κορυφής για τις γυναίκες στην, σε τομείς τεχνολογίας. Ε, έχουν γίνει πολλά, αλλά βεβαίως τα προβλήματα δεν, δεν είναι λίγα. Η συμφιλίωση, ας πούμε, της επαγγελματική και της προσωπικής ζωής. Η νομοθεσία σχετικά πρέπει να τροποποιηθεί για να ενθαρρύνει, για να διευκολύνει τους ε, εργοδότες ώστε να μπορούν να κάνουν περισσότερα για να παρέχουν ε, ε, προστασία στις γυναίκες, βοήθεια ό,τι αφορά την φύλαξη των παιδιών τους και επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα. Η μάχη αυτή δεν σταματά. Εξεκολουθούμε να μην έχουμε πολλά κορίτσια που σπουδάζουν σε τεχνολογικούς κλάδους ή σε φυσικές επιστήμες. Και βεβαίως υπάρχει και ε, το μισθολογικό κενό. Το ίδιος μισθός για την ίδια δουλειά εξακολουθεί να παραμένει ένα όνειρο. Ευχαριστώ κυρία Μπόροβιτς από τη Γαλλία, η κυρία Μαρή Πιέρ Ριξόν. Ευχαριστώ. Στην Γαλλία, όπως πολλές από εσάς, αντιμετωπίζουμε ένα διτό πρόβλημα. Πρώτον, μεταξύ της δεκαετίας του 80 και του 90 στην Γαλλία υπήρχαν 40 έως 50% γυναίκες στο χώρο της ψηφιακής ε, τεχνολογίας και της ε, επικοινωνίας. Τώρα είναι 27%, 19% της ψηφιακής εταιρείας. Επίσης, κάτι που είπατε τώρα, σε 10 με 15 χρόνια, ε, ε, τα επαγγέλματα που είναι σε ε, φάση σύμβασης θα έχουν γίνει ψηφιακά. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και επίσης ε, θα υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, ιδίως στην ιατρική, από την τεχνητή ευθεία και την ρομποτική. Πολύ σύντομα οι διαγνώσεις δεν θα βγαίνουν μόνο από επαγγελματίες του χώρου υγείας, αλλά και από λογισμικά. Λογισμικά που δεν θα διέπονται μόνο από σεξιστικά στερεότυπα, αλλά θα έχουν και εφαρμογές για να καθορίζουν τη γυναικεία υγεία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό για τη σωματική ακόμη υγεία των γυναικών. Τώρα, στο Εθνικό Συμβούλιο το οποίο προεδρεύω, αποφασίστηκε να συνταχθεί έκθεση και μιλάμε με ερευνητές, μελετητές, κοινωνιολόγους, επιχειρηματίες και πρόεδρους εταιριών, ε, γιατί όλοι επισημαίνουν τα εξής το πρώτο είναι ότι υπάρχουν τα στερεότυπα, αυτές οι προκαταλήψεις που τις έχετε ήδη αναφέρει και μετά υπάρχει ο σεξισμός στον τομέα των ψηφιακών εταιριών είναι σημαντικό να το ε, υπενθυμίζουμε, διότι δεν αρκεί μόνο οι γυναίκες να έχουν υπόψη τους ε, την έλλειψη γυναικών στον χώρο των εταιριών αυτών, αλλά είναι και ευθύνη συλλογική, είναι ευθύνη όλων μας. Πρέπει να θυμάται ο χώρος των ψηφιακών εταιριών ότι δεν ε, υποδέχεται αρκετές γυναίκες όπως άντρες. Και σε κάποιες σχολές ε, που προετοιμάζουν για τα ψηφιακά επαγγέλματα, ε, σχολές ε, που πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν σκεφτεί να προβλέψουν λόγου χάρη γυναικείες τουαλέτες στις εγκαταστάσεις τους πριν από μερικά χρόνια. Αυτό γιατί ήταν ελάχιστος ο αριθμός γυναικών που έφταναν ως εκεί. Και τελευταία παρατήρηση, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω μια προσωπική μου εμπειρία. Την περασμένη μόλις εβδομάδα οργάνωσα συνεδρίαση στην εκλογική μου περιφέρεια με συμμετοχή μαθητών και φρόντισα να έρθουν ερευνήτριε που ασχολούνται με θέματα κρυπτογράφηση και τεχνητής ευφυΐας. Και μια μικρή μου είπε Είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά. Ε, και αυτό που ήθελα να σας πω είναι η μαρτυρία αυτών των κοριτσιών και γυναικών ε, γιατί ανησυχούν για το μέλλον τους. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμη δύο ομιλητές, αλλά θα παρακαλέσω τον Μάτι Τουρινέλ από τη Φιλανδία και τον Νικόλ από την Γερμανία να μιλήσουν μόνο ένα λεπτό, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ε, Πρώτα ο κύριο Τόρβινεν από τη Φιλανδία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλες τις γυναίκες του κόσμου που κάνουν αυτόν τον κόσμο ένα πολύ ευχάριστο μέρος να ζει κανείς. Μάτι Τόρβινεν ονομάζομαι από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Για το... Είμαι μέλος του κόμματος της μπλε μεταρρύθμισης. Ε, εκτιμώ το ότι θίγεται τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα για την υποεκπροσώπηση των, γυναικών στον τομέα της ε, πληροφορικής και σε άλλους τεχνικούς κλάδους, ακόμα και σε χώρες ε, που είναι πολύ διάσημες για την ισότητα μεταξύ των φίλων, όπως είναι η Φιλανδία. Όλοι πρέπει να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να μπουν στον προγραμματισμό, να μπουν στις, ε, στα, στον μηχανικό κλάδο, στους τεχνολογικούς κλάδους, γιατί υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανισορροπία ανδρών και γυναικών σε αυτούς τους κλάδους. Αν ε, διατηρήσουμε τα στερεότυπα που υπάρχουν ότι η πληροφορική είναι για τους άντρες, τότε θα χάσουμε το τεράστιο δυναμικό και τις ιδέες που μπορούν να προσφέρουν οι γυναίκες στον ε, τομέα αυτό. Εγώ είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα και βλέπω πραγματικά πόσο μεγάλο δυναμικό υπάρχει σε ό,τι αφορά την καινοτομία και πώς οι γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό ο προγραμματισμός και η πληροφορική θα πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία, σε αγόρια και σε κορίτσια εξίσου, για να μπορέσουμε να έχουμε στο τέλος περισσότερα κορίτσια που θα αποφασίσουν τελικά να ακολουθήσουν μια τεχνολογική καριέρα. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι περισσότερη διεθνή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων στον κλάδο της πληροφορικής, έτσι ώστε αυτός ο κλάδος να διαφημιστεί ακόμη περισσότερο, να γίνει ακόμη πιο ελκυστικός. Η Ελίντα Λιούκα έχει γράψει ένα παιδικό βιβλίο, είναι μια γνωστή συγγραφέα και έχει γράψει ένα παιδικό βιβλίο για την πληροφορική ακριβώ. και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά προσπαθώντας να προωθήσει την πληροφορική μεταξύ των κοριτσιών. Οι γυναίκες έχουν πραγματικά τεράστιες δυνατότητες για την πληροφορική και το φύλλο δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο όταν διαλέγει κανείς μια τεχνολογική ή καριέρα πληροφορικής, όπου και να βρίσκεται στον κόσμο. Να ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο της Γερμανίας. Ναι, ευχαριστώ. Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ όλες τις γυναίκες που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών και μετά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ακούστηκε ότι θα κρατήσει άλλα 100 χρόνια μέχρι να πετύχουμε την απόλυτη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα αυτό και αυτό που μου αρέσει είναι αυτό που ακούστηκε σήμερα, ότι οι γυναίκες χρειάζονται πρότυπα. Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, δουλεύω 8 χρόνια στην, δούλευα 8 χρόνια στην Γερμανία σε αυτόν τον κλάδο πριν μπω στην πολιτική. Και αυτό που διαπίστωσα είναι ότι η συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής δεν είναι δεδομένη. Οι γυναίκες εξακολουθούν να, είναι, ε, να εκπροσωπούνται μερικώς σε θέσεις ευθύνες. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε ευκαιρίες ψηφιοποίησης στις γυναίκες, να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές που υπάρχουν για να βοηθήσουμε να, δημιουργούν, να δημιουργηθούν νέα εργασιακά μοντέλα αλλά και κυρίως να προωθήσουμε τις ε, περιοχές της υπαίθρου, γιατί αυτές είναι ακριβώς που ε, αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και το μισό από, τον, το, από τους πολίτες της Ευρώπης ζουν στην Ήπεθρο και πραγματικά εκεί υπάρχει τεράστια ανάγκη για να, πάμε πολύ, για να κάνουμε περισσότερη πρόοδο. Επίσης, αυτό το, αυτή η κίνηση προς τα πίσω που βλέπουμε πολλές φορές από κόμματα πολιτικά για την θέση των γυναικών στην οικογένεια μόνο και στο σπίτι μόνο. Πολλοί είναι αρκετά πετυχημένοι σε αυτό και γι' αυτό πραγματικά είναι κρίμα. Πρέπει όλοι να σταθούμε απέναντι σε αυτό έτσι ώστε να μην ε, προχωρήσει κι άλλο. Ευχαριστώ. Κλείσαμε λοιπόν τον ε, κατάλογο των ομιλητών και τώρα να κάνουμε μία μικρή περίληψη δίνοντας πρώτα το λόγο για να ακούσουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα να δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις στα πρώτα δύο, σύμφωνα με τα στατιστικά. Το πρώτο ερώτημα ήταν ποιες μεταξύ των τεσσάρων χωρών ε, κρατών μελών έχουν την υψηλότερη ε, ε, προσώπηση στην πληροφορική. Η Βουλγαρία λέγεται ότι είναι 28% ειδικών περιπληροφορικής, το υψηλότερο μάλιστα ποσοστό στην Ευρώπη, συγχαρητήρα στη Βουλγαρία. Απάντηση στη δεύτερη ερώτηση Κατά την άποψή σας, ποιο είναι, ποια είναι το ποσοστό των ε, αποφύτων πληροφορικής γυναικών. 17 είναι η σωστή απάντηση. Και μόνο 10% αυτού του 17% των αποφύτων συνεχίζουν ε, την ε, σταδιοδρομία τους στον κλάδο της πληροφορικής. Οπότε διπλά αρνητικό το φαινόμενο. μετά, η πιο δημοφιλής ερώτηση που μπήκε μέσω του σλάιντο είναι πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τους άντρες στην επίτευξη της ισότητας των φύλων. Και θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την κυρία Επίτροπο σύντομα να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά και από το κοινό και από το διαδίκτυο. Έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω όλες τις παρεμβάσεις για τις οποίες σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου μια φράση. Το θέμα είναι να δώσουμε παραδείγματα και αυτά να ε, μπορέσουν να εκφράσουν και ένα μήνυμα. Σήμερα, για να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, πρέπει να έχουμε υπόψη και τις εκφράσεις και μορφές βίας με τις οποίες μας φέρνουν αντιμέτωπους καθημερινά τα μέσα της ψηφιακής τεχνολογίας θα πρέπει οι γυναίκες να προετοιμαστούν για να μπορέσουν να χειριστούν τις νέες τεχνολογίες και στον χώρο της εκπαίδευσης και μετά στην αγορά εργασίας. Εδώ απαιτούνται κοινέ προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα παραδείγματα καλών πρακτικών που μας δώσατε. Ακριβώς αυτό χρειάζεται, να τα διαδώσουμε, να τα προβάλλουμε. Και έτσι μόνο θα έχουμε περισσότερη ε, επιτυχία στα ICT, στην Ισπανία, την Πολωνία, την Γερμανία. Με συγχωρείτε αν κάποιον τον ξέχασα, αλλά προφανώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, τους κινδύνους του, του ψηφιακού κλάδου. Προσφέρει ευκαιρίε, αλλά απειλεί κιόλα με περισσότερη φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, από περιθωριοποίηση κάποιων ολόκληρων περιοχών. Να δούμε τι συμβαίνει Ε, με την ε, διασύνδεση αυτή τη στιγμή, 76% των οικοκυριών σε αστικέ περιοχέ είναι καλά συνδεδεμένα ή τρίω καλά συνδεδεμένα, 40% είναι το ίδιο ποσοστό στην Ήπεθρο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να μην ξεχνάμε ότι και οι άντρε μπορούν να γίνουν πρέσβει και αγγελεφόροι του μηνύματός μα. Από τον Φεβρουάριο ξεκινήσαμε μια ενημερωτική εκστρατεία που ονομάζεται Safer Internet for EU, ασφαλέστερο διαδίκτυο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο το 2018 θα οργανώσουμε δράσει σε όλα τα κράτη-μέλη ε, με πρέσβεις, ε, αυτούς που μεταφέρουν το μήνυμά μας, να μπορούν να μας υποστηρίξουν εφόσον το θέλουν, για την απαραίτητη εκπαίδευση και καλλιέργεια που απαιτείται, για την καλή χρήση του διαδικτύου, του ίντερνετ, ε, για την κύβερνο ασφαλειά μας, για να εξηγήσουμε στους νέους ότι στον κόσμο του διαδικτύου υπάρχουν ίδιες αξίες, ίδια ελευθερία, δυνατότητες και απειλές, όπως στον κανονικό κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμά μου σήμερα και εγώ εύχομαι να έχουμε όλο ένα και περισσότερου συνεργάτε. Ο τελευταίο ε, ε άντρα που ήρθε να ενωθεί στι προσπάθειέ μα είναι ο Βιμ Βάντερ. είναι πραγματικά ε, ένα καλό πρότυπο, είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να μα δώσει και αυτό πρέπει και στα σχολεία να το προβάλλουμε και να το διαδώσουμε. Να ξέρουν οι νέοι τι μπορούμε να κάνουμε και ότι επιζητούμε θετικά αποτελέσματα και ποιότητα. Ε, θα λάβω πολύ σοβαρά και τη σύσταση για την ε, φωνή της Ευρώπης και τη θέση των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ και την κυρία Εστρέλα για τις ε, ευχές της. Χαρήκαμε πολύ που σας ξαναείδαμε. Ε, λίγες εκθέσεις έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο που έχουμε τόσο πολλούς λόγους να θυμόμαστε. Μια από αυτές είναι η έκθεση Εστρέλα που σημάδεψαν την ε, πορεία του Ευρωκοινοβουλίου. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να συνεχίσουμε αυτή την πορεία να δώσουμε το καλό παράδειγμα με την σωστή προβολή. Οι γυναίκες που έχουν δυνατότητες, δεξιότητες και προσόντα είναι σήμερα εδώ έχουν ε, τα χαρτιά στα χέρια τους, αλλά πρέπει να τις προλάβουμε, μας είπα, να τις προβάλλουμε. Μας είπατε τώρα ότι μιλήσατε εσείς τις προάλλες με γυναίκες ειδικές στην κρυπτογράφηση και την τεχνητή ευθεία. Τις ξέρουμε, πρέπει όμως να τις φέρουμε στο προσκήνιο. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσω και την ε, εφαρμογή της στατικικής για να υπάρχει λίγη περισσότερη συνοχή μεταξύ των διαφορετικών δράσεων. Και πάλι το βασικό μήνυμα από μένα είναι δράση, πράξη σε όλα τα επίπεδα. Εάν δράσουμε σε αυτό το μέτωπο, όχι μόνο άντρε, γυναίκες αλλά και άντρες, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, όλοι μπορούμε κάτι να συμβάλλουμε. Έστω και ένα πετραδάκι και έτσι θα, ε, ένα λιθαράκι μάλλον και έτσι θα πετύχουμε να επιτεθεί δροματική πρόοδο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλους, σας εύχομαι καλή δύναμη ε, και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η μέρα πρέπει να γιορτάζει 365 μέρες το χρόνο και όχι μόνο μία. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Τώρα τρία λεπτά στην κυρία Παραντίκα από το Άλτε για κάποια τελικά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και βέβαια ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Και εγώ χαιρετίζω εδώ όλος ιδιαίτερος την παρουσία της κυρίας Εστρέλα η οποία αγωνίστηκε τόσο πολύ με τις εκθέσεις της και πράγματι άφησε και εκείνη ένα μέρος της καρδιάς της εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνουμε πολλά. Έχω την αίσθηση ότι βαρεθήκαμε να ακούμε τέτοια και τα ίδια. Είμαι πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έχουμε πάνω από το 61% πτυχιούχων πανεπιστημίου. Δεν είμαστε όμως τα διοικητικά συμβούλια, δεν είμαστε σε θέση αποφασής. Ε, υποφέρουμε από την ε, βία σε βάρος των γυναικών. Ε, τα είπε και η Επίτροπος από τις μελέτες που έχουν γίνει και τα νούμερα που έχουμε για τη βία, την ενδοικογενειακή βία ή τη σεξουαλική παρενόχληση είναι φοβερά. Τα στερεότυπα παραμένουν. Και χτες το είδαμε αυτό και σήμερα το πρωί. Δεν συμμετέχουμε αρκετά στα μέσα ενημέρωσης. Τι συμβαίνει, γιατί στις ε, τεχνολογίες, στην πληροφορική, γιατί ε, ακριβώς επειδή υπάρχουν τα στερεότυπα, ισχύει και εκεί το ίδιο. Τι είναι οι τεχνολογίε πληροφορικής, αποτελούν μια ευκαιρία, αλλά αποτελούν και μια ανάγκη. Το είπε η Επίτροπος, αποτελούν ευκαιρία γιατί ε, θα τις χρειαστούμε όλο και περισσότερο τις θέσεις απασχόληση σε αυτό το κλάδο, αυτές τις δεξιότητες δηλαδή, για να αναπτυχθεί ο οικονομικός κόσμος, για να προχωρήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Αποτελεί όμως και ευκαιρία για την ύπεθρο. Και εμείς αυτό το υπογραμμίζουμε σε έκθεση που εγκρίθηκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα υποβάλουμε για την 62η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και εκεί υπογραμμίζουμε ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί μέσο για να αντιμετωπιστεί η ανισότητα και η φτώχεια. Τι γίνεται όμως, χρειάζονται επαγγελματίες, γυναίκες και όλες οι μελέτες μας λένε ότι παντού όπου συμμετέχουν οι γυναίκες και στην πληροφορική δηλαδή οδηγούν σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Υπάρχει περισσότερη δημιουργικότητα, επιχειρήσει εκεί δουλεύουν καλύτερα και μάλιστα χρησιμοποιούν και καλύτερα και του οικονομικού πόρου εκεί. Οπότε γιατί Είμαστε περισσότερες γυναίκες, έχουμε τόσα θετικά, παρόλα αυτά δεν τα καταφέρνουμε. Και στις τεχνολογίες πληροφορικής από ό,τι φαίνεται μειώνεται και η παρουσία μας. Οι εκστρατείες, ναι, συμφωνώ με την εκστρατεία ε, που λέει αν δεν υπάρχουν γυναίκες να μην υπάρχουν ούτε και πάνελ. Η, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στη Μαδρίτη έκανε μια πρωτοβουλία την προηγούμενη εβδομάδα και συμφωνήσαμε και εμείς ότι με τέτοιες εκστρατείες μπορούμε να πετύχουμε πολλά αλλά πρέπει να κάνουμε και περισσότερο. Πρέπει να υπάρχει δέσμευση από όλου υπέρ νομοθεσίας, δεσμευτικής όμως, υποχρεωτική. Το 2005 στη χώρα των Βάσκων εγκρίθηκε ένας νόμος για την ισότητα που έκανε υποχρεωτικές τις ποσοστώσεις και ο πρόεδρος είπε ότι αυτός ο νόμος ήταν ο πιο σημαντικός της θητείας του. Και τώρα η χώρα των Βάσκων είναι σαν ένα μικρό εργαστήριο με παρουσία των γυναικών και στην πολιτική ζωή αλλά και αλλού πάρα πολύ σημαντική. Κοιτάξτε το, δεν λέω ότι τα πετύχαμε όλα γιατί η ισότητα δεν είναι μία κατάκτηση που δεν υπάρχει περίπτωση να πάει πίσω. Λοιπόν, χρειάζεται προβολή των γυναικών. Αλλά γι' αυτό οι γυναίκες πρέπει να είμαστε αποφασισμένες να αναλάβουμε ηγετικούς ρόλους, να στηρίξουμε τις αξίες μας που είναι πολύ σημαντικές και να μην μιμούμεθα τους άντρες για να αναγνωριστούμε. Ο αγώνας λοιπόν είναι υπόθεση όλων. Πάντως για να πετύχουμε αυτή την εμπιστοσύνη στις γυναίκες πρέπει να συνεργαστούμε γιατί τα μέτρα πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Μην χάνουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μπαραντίκα, ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ και όλους τους συμμετέχοντες στην διάσκεψη αυτή. Το επόμενο πάνελ θα το αναλάβει άλλη συνάδελφος. Παρακαλώ, ελπίζω να είσαστε καλύτεροι στη διανομή του χρόνου από μένα. Thank you very much and also warm welcome from... Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε και από μένα. Δεν θα κάνουμε κανένα διάλειμμα γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε δυστυχώς, οπότε κατευθείαν περνούμε στο τρίτο πάνελ. Ήδη έχετε συζητήσει το ρόλο των γυναικών στα ΜΜΕ και το θέμα της ψηφιακή ε, συμπερίληψης και της ισότητας των φύλων. Και τώρα πάμε στην τρίτη συζήτηση που έχουμε προβλέψει για σήμερα, που θα διαχειριστεί ένα πολύ σημαντικό θέμα και πολύ σημαντικές εξελίξεις που είδαμε να υπάρχουν, γιατί ο ψηφιακός κόσμος χρησιμοποιείται και από φεμινιστές και από εκπροσώπους των δικαιωμάτων των γυναικών τα τελευταία χρόνια για να αγωνιστούν για τα δικαιώματα των γυναικών, για την ε, ισότητα σε όλο τον κόσμο και θέλουμε να ακούσουμε ακριβώς αυτά τα κινήματα και να τα συζητήσουμε. Γι' αυτό έχουμε καλέσει την Dagmar Schumacher, που είναι η επικεφαλής του Γραφείου των Βρυξελών του ΟΗΕ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται στον τομέα αυτό και βεβαίως μετά θα ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον τα δικά σας σχόλια και τι γίνεται στις δικές σας χώρες και τι είδους συζητήσεις γίνονται στις δικές σας χώρες και τι προσπαθούν να κάνουν οι εκπρόσωποι των διαφόρων σωματείων που μάχονται για τα δικαιώματα των γυναικών. Πριν ξεκινήσουμε από την παρουσίαση της κυρίας Σουμάχερ θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι το slide για να σας ε, θέσουμε κάποια ερωτήματα. Δύο ερωτήματα και πάλι και παρακαλώ να τα απαντήσετε. Θέλουμε να μας πείτε αν ξέρετε και πόσα ξέρετε για τα διάφορα ψηφιακά κινήματα που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που θέλουμε να σας θέσουμε είναι το εξής. Πόσες από αυτές τις ε, γυναίκες ε, γνωρίζετε που είναι επικεφαλής διαφόρων κινημάτων, οργανώσεων ε, μέσω της, ε, των ΜΜΕ. Πρώτη, Αλίσα Μιλάνο, ε, Μπάρμπαρα Νοβάτσκα. Τρίτη ομάδα, Αλίσια Γκάρσα, Πατρίς Κουλόρς και ο Παλτομέτη, Η Σέριλ Σάντμπεργκ, Ρέιτσελ Σκλάρ, η Μαλάλα Ιωσαυζάη. Και μετά έχετε και την επιλογή να πείτε ότι δεν ξέρω καμία από αυτές τις γυναίκες. να σας δώσω κάποια δευτερόλεπτα για να δείτε το ερώτημα και να το απαντήσετε, αλλά βεβαίως έχετε τη δυνατότητα για τη διάρκεια της συζήτησης να δώσετε την απάντησή σας. Μπορείτε απλώς να μπείτε στην ιστοσελίδα του Slido και ε, να βάλετε τον κωδικό IWD 2018 και μετά μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτά τα ερώτηματα. Δεύτερο ερώτημα πρέπει να κάνετε μια εκτίμηση. Πόσοι χρήστε του Facebook και του Twitter έχουν απαντήσει στην ε, ε, ε, εκστρατεία MeToo εντό των πρώτων 48 ώρων μετά το tweet της Αλίσσα Μιλάνο. Πόσοι άνθρωποι πιστεύετε ότι απήντησαν εντό των πρώτων δύο ημερών. 100.000 άνθρωποι, 500.000 1.200.000 ή 5.700.000 και σε αυτό το ερώτημα. Κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης θα έχετε την, ε, το χρόνο να απαντήσετε και βεβαίως περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τις απαντήσεις σας. Και τώρα, επειδή δεν έχουμε χρόνο πολύ, θα δώσω αμέσω το λόγο στην κυρία Ντάγμαρ Σουμάχερ για να μας δώσει τη δική τη ε, άποψη για το τι γίνεται στην, ε, στο ψηφιακό τομέα και τα διάφορα κινήματα των γυναικών και τι πρέπει να προσέξουμε. Και ίσως να μας πει και λίγα πράγματα για το ποιε είναι οι προκλήσεις. Ευχαριστώ Τέρι, ευχαριστώ και την Επιτροπή ε, Γυναικών για την πρόσκληση και που έβαλε το πολύ σημαντικό αυτό θέμα στην σημερινή ημερήσια διάταξη. Βλέπουμε πραγματικά τεράστια κινητοποίηση για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Ξέρουν οι πολίτε ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι σημαντικά θέματα, είναι θέματα καθημερινά, διεθνή και εθνικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τη επίμονη κινητοποίηση των γυναικών και των κινημάτων των γυναικών που πιέζουν για αλλαγή και που θέλουν να λογοδοτούν οι κυβερνήσει. Σήμερα τα κινήματα αυτά βασίζονται στις υπάρχουσες ψηφιακές τεχνολογίες και στα κοινωνικά δίκτυα που αποτελούν τους καταλήτες για αυτά τα κινήματα. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή, για την ενημέρωση, την πρόσβαση, την κινητοποίηση, την υπεράσπιση, την οργάνωση ε, ε, διαφόρων ε, εκδηλώσεων κλπ. Αν δούμε τις, τους διάφορους κόμβους που υπάρχουν μεταξύ των κινημάτων των γενικών και της ψηφιοποίηση και πώς το γράμμα όλων αυτών διαμορφώνει και το πνεύμα των κινημάτων. Η ελληνική και μέσω των ε, ε, ε, εκδηλώσεων στα, κοινωνικά δίκτυα οι πολίτες μπορούν να προωθήσουν την ισότητα των φύλων. Κάποια από τα κινήματα αυτά έχουν βρεθεί και στους επιχείρους τίτλους των εφημερίδων, κάποιοι κινούνται στις κουίντες. Προσπαθούμε λοιπόν όλοι να κινητοποιήσουμε την, ε, τα κινήματα αυτά και να βελτιώσουμε την επιρροή και σε νομοθετικό αλλά και σε επίπεδο κοινωνικών μεταρρυθμίσεων μέσω της ε, πάυσης της ε, βίας στον χώρο εργασίας, πρόσβαση στις υπηρεσίες, καλύτερη προστασία των μεταναστών και προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε τους πάντες σε αυτά τα κινήματα. Στην ε, Διεθνή ημέρα των ε, γυναικών ξέρουμε ότι ε, πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο μείγμα φωνών, αλλά πολύ ε, πολλές γυναίκες σε όλο, τον κόσμο παραμένουν σιωπηρές. Πρέπει λοιπόν να, να υπάρξει η στιγμή που θα αλλάξουν τα πράγματα, να πάψει η ασυλία και ο κύκλος αυτών των, ε, γυναικών που μένουν εκτός των πάντων, κυρίως αν ζουν στις, ε, στην Ήπεθρο. Ε, Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αλλαγή, κυρίως για αυτούς που την έχουν ανάγκη περισσότερο. Τα κοινωνικά μέσα έχουν δώσει στις γυναίκες την δυνατότητα να ανθίσουν πραγματικά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων σκανδάλων, οι γυναίκε χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά δίκτυα για να κατηγορήσουν όσου του παρενοχλούν σεξουαλικά και να καταδείξουν περιστατικά βία πολιτικοί ε, ηγέτες, ε, εταιρείε θεωρούνται πλέον υπόλογοι για τα προβλήματα που ε, δημιούργησαν. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πίεση για τα στανότερα στρώματα των, της κοινωνίας μας και οι πολίτες μπορούν να κάνουν πραγματικά την αλλαγή, κυρίως ό,τι φορά την απόκτηση ισότητας μεταξύ των φίλων. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και το hashtag για τη συζήτηση αυτή που κάνει πάρα πολύ εύκολη τη συμμετοχή όλων στην αλλαγή που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Βοηθά πραγματικά να έρθουν στο φω όλα αυτά τα ζητήματα που μα απασχολούν. Οι στόχοι τη βιώσιμη ανάπτυξη τη ε, του θεματολογίου για το 2030 και κυρίω οι στόχοι που σχετίζονται με τι γυναίκε και την τεχνολογία παρέχουν μια ιστορική ευκαιρία για να ανατρέψουμε τι ε, ανισότητε στον τομέα τη ε, ψηφιακής τεχνολογία και να μετατρέψουμε τα λόγια σε πραγματικέ δράσει. Παρ' όλα αυτά, χωρί να υπάρχει κλιμάκωση τη πολιτική αλλά και των επενδύσεων, υπάρχει κίνδυνο, τεχνολογικέ αλλαγέ αλλαγές να συνεχίσουν να ενισχύουν τις υπάρχουσες ανισότητες. Γι' αυτό, αν ε, θέλετε, μπορώ να σας δώσω και κάποια α, παραδείγματα. Παρακαλώ, δεν θα σας πω πολλά, οπότε κάντε λίγη υπομονή. Ήδη μιλήσαμε για το κίνημα μητού και επειδή ακριβώς το θέμα είναι και το ερώτημα που έχουμε θέσει είναι για το μητού, δεν θα πω πολλά, αλλά θα πω απλώς ότι οι γυναίκες έχουν την πλατφόρμα για να μπορούν να βγουν στο φως και να δουν πόσες ακόμα γυναίκες είχαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια περιστατικά σεξουαλικής βίας. Δεύτερον, η Sheryl Sandberg έχει ξεκινήσει το δικό της hashtag για να βοηθήσει την ε, ανάληψη ε, θέσεων ηγεσίας από τα κορίτσια. Είχαμε τα pink sticks που είναι μια εξατία που ε, στοχεύει τα, τα προϊόντα που η βιομηχανία θεωρεί ως στερεοτυπικά γυναικεία. Και αυτό συνδέεται και με γενικότερα τα στερεότυπα που υπάρχουν. Θέλουμε να, να αλλάξει το τι γίνεται στη βιομηχανία διαφημιστική και θέλουμε βεβαίως και τους άντρες στο πλευρό μας. Από την πολιτική του πτυχή είδαμε στην Αραβική Άνοιξη και στο κίνημα στην Αίγυπτο με την ε, χειραφέτηση των γυναικών. Το τι έγινε όταν ξεκίνησαν όλα αυτά ήδη από το 2010. Ήδη το 2011 ξεκινήσαμε αντίστοιχε εξαρτίε για να αντιμετωπίσουμε την ε, σεξουαλική παρενόχληση στην Αίγυπτο μέσω μια ε, δυνατότητα online κατα, καταγγελία και μέσω SMS. Υπάρχει το hashtag Bring Back Our Girls από την Ιγυρία για την Boko Haram και νομίζω ότι θυμάστε τι εξαρτίε που έγιναν για τα κορίτσια αυτά, γιατί πραγματικά δεν έχουμε φτάσει στο στόχο μας ούτε εκεί. Έχουμε το Shady Sites με, με ιστοσελίδες που ε, στοχεύουν γυναίκες. Έχουμε το 2017 το hashtag Women's March που ε, συνδύασε πραγματικά πολλά κινήματα αντίδρασης σε όλες τις ε, υπήρους. Είχαμε την, ε, πολλές εκστρατείες, το Time's Up και άλλες. Spotlight and Violence επίσης, άλλο hashtag από την ε, πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αντιμετωπιστεί η βία κατά των γυναικών παγκοσμίω. Επίσης σήμερα έχουμε και για, τη δική μας, για το δικό μας τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας ένα νέο hashtag που ονομάζεται Time is now. Τώρα είναι η ώρα για να δημιουργήσουμε αυτό το κίνημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι αύριο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και πρέπει να συμπεριλάβουμε και του άντρε σε αυτό το πολύ σημαντικό πλαίσιο. Και το άκουσα αυτό να λέγεται και από την προηγούμενη σύνοδο. Το H4C επίση είναι μια εξαρτία που μπορεί να βοηθήσει για να επιτύχουμε την ισότητα των φίλων. Επίσης, ως ε, γυναίκες στον ΟΗΕ έχουμε ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα για διαφορετικά ορόσημα για την ισότητα των φύλων που μόλις δημοσιεύθηκε. Και σας ενθαρρύνω να το δείτε. Στο τέλος υπάρχει το τελευταίο, το πιο πρόσφατο ορόσημο που έχει να κάνει με τον ψηφιακό ακτιβισμό. Και αυτό είναι ακριβώς για το, το θέμα για το οποίο μιλούμε και θέλουμε να προωθήσουμε. Ο ψηφιακός ακτιβισμός που βεβαίως πρέπει να υποστηρίξει το τι γίνεται και offline. Και εδώ μπορώ να έρθω στις προκλήσεις όπως με είπε Τέρι. Καταρχάς, οι γυναίκες πολύ συχνά δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στο ίντερνετ όπως οι άντρες. Επίσης και σήμερα το πρωί το ακούσαμε αυτό, οπότε δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα αν όλε αυτέ οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε δεν ε, ε, αντιμετωπιστούν και στα πλαίσια του ψηφιακού ακτιβισμού. Βεβαίω πρέπει να συμμετάσχουμε περισσότερο online και ίσως να πρέπει να είμαστε λιγότερο ενεργές offline. Πρέπει να, να τηρήσουμε την πίεση και στα δύο μέτωπα. Και επίσης κλείνοντας να πω ότι βεβαίως γενικώ η καινοτομία και η ατζέντα της, αλλά και η πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στον ε, κλάδο της πληροφορικής έχει τεράστιο δυναμικό, κυρίως ό,τι αφορά την πρόσβαση στην πληροφόρηση, σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της εκπαίδευση, τι εμπορικέ ευκαιρίε, την πρόσβαση τη αντίστοιχη υπηρεσίας και την οικονομική ανεξαρτησία. Και πάνω απ' όλα την ε, πρόθεση του κινήματο για την ισότητα των φύλων. Πρέπει να αμβλύνουμε τι φωνέ των γυναικών και το κίνημα πραγματικά είναι ε, όριμο, ο χρόνο είναι όριμο για να γίνει αυτό. Και θα ήθελα να ακούσω τι δικέ σα προτάσει, τι δικέ σα ιδέε και σα εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη Διεθνή ε, ημέρα για, την για τα δικαιώματα των γυναικών. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τόσο καλή αφορμή για να ξεκινήσει η συζήτηση. Αναφέρατε δύο πολύ ισχυρά κινήματα που έχουν φέρει αλλαγή στην κοινωνία μας τους τελευταίους μήνες και χρόνια. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε βουλευτές για να θέσουν ερωτήσεις και να κάνουν τα σχολεία τους. Πρώτη ομιλήτρια από την Πορτογαλία, η Χερμάνα Ρόχα. Ρόζα. Ε, ευχαριστώ ε, καταρχάς ήθελα να υπογραμμίσω ότι η συζήτηση αυτή έχει μεγάλη σημασία για την Πορτογαλία και είναι πολύ επίκαιρο για την Ευρώπη και το διεθνές προσκήνιο. Θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο ο ρόλος και η σημασία των νέων τεχνολογιών στα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης, καθώς και το πώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών. Οι τεχνολογίες, ιδίως οι τεχνολογίες ενημέρωσης και επικοινωνίας, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μεταμόρφωση του κοινωνικού πολιτισμού πολιτικού και οικονομικού βίου σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα είναι ένα τρόπο να προωθηθούν ευκαιρίε ώστε άντρε και γυναίκε να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή και παραγωγική εργασία. Ωστόσο, πέραν από την θετική εξέλιξη των ποσοστών απασχόληση επαγγελματιών ε, ε, από το τι σχολές επικοινωνίας και πληροφόρησης, πληροφορική. την τελευταία δεκαετία βλέπουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλύπτονται όλες οι ανάγκες του κλάδου και κυρίως από γυναίκες. Εδώ υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της ζήτηση και την προσφορά ειδικών ICT στην Ευρώπη, ιδίω γυναικών, και βάσει της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Ιανουάριο του 2014 εκτιμάται ότι το 2020 το χάσμα αυτό θα είναι 900.000 ε, θέσεις και θα παραμένουν κενές. Ε, γιατί λείπουν οι απαραίτητε δεξιότητε. Σκεφτείτε τι συμβαίνει όταν μιλάμε για γυναίκε στον χώρο των ICT. Στις, στην Πορτογαλία στι ICT οι γυναίκε είναι ελάχιστα εκπροσωπούμενε, είτε στον τομέα τη εκπαίδευση είτε τη εργασία. Το 2016 στην Πορτογαλία οι γυναίκε που ασχολούνται με τον τομέα αυτό ήταν 59%, αλλά μόλι 33% ε, ε, στον τομέα τη μηχανική, των πολυτεχνείων. Επίση, στον τομέα τη εκπαίδευση 82%, ενώ στον τομέα τη υγεία και τη κοινωνική κοινωνική προστασία 67%. 77% συγγνώμη. Επίση για, τη για την δημόσια διοίκηση και τι επιχειρήσει, μόνο 56% ήταν οι θέσει που καλύπτονταν από τι γυναίκε. Ε, εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε κατά πόσο οι γυναίκες παραμένουν μειονότητα στον ε, ε, στους κλάδους αυτούς και στους μισθούς και στις θέσεις που καλύπτουν. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλυφθούν αυτά τα κενά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερη από τις κάτω χώρες, η κυρία Τίλα. Εκτός μικροφώνου η Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και ευχαριστούμε που ε, μας παρουσιάζετε το έργο σας. Ε, πολύ καλό παράδειγμα προς μίμηση και ελπίζω να βρούμε και ευρωπαϊκά ανάλογα παραδείγματα σε κάποιο καιρό. Και ε, καλά κάνατε και αναφέρατε την Λίγκο ως την Λέγκο ως παράδειγμα για γυναικεία πρότυπα που προωθούνται με τις γυναίκες αστροναύτες λόγου χάρη που εργάστηκαν στην Άσα. Ε, και τα πέντε σχετικά κουκλάκια που έχουν ε, προταθεί. Μιλάμε σήμερα το πρωί για την καταπολέμηση των στερεοτύπων. Όμω τα στερεότυπα δεν μπορεί απλώ να εξαλειφθούν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και είναι εφικτό είναι να προσθέσουμε θετικά στερεότυπα και να τα αξιοποιήσουμε. Ιδίω στον χώρο των ψηφιακών ε, εξελίξεων. Διότι οι γυναίκε έχουν χάρισμα στην επικοινωνία. Είναι στερεότυπο και είναι και θετικό. Οι γυναίκε είναι έξυπνε και ευθύ. Οι γυναίκε ε, είναι και αναζητούν τα υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Εργάζονται καλά σε ομάδα. Μπορούν να επικοινωνήσουν, ε, να δημιουργήσουν και να κερδίσουν την αποδοχή. Αυτά τα στερεότυπα μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερο θετική αποτίμηση. Εδώ λοιπόν πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με, με τους άντρες και να φροντίσουμε από κοινού να επιδιώξουμε να ψώσουμε φωνή η οποία είναι και δυνατή. Μιλώντας για φωνή, αναφέρατε κάποια παραδείγματα από την ψηφιακή επανάσταση για να την πω έτσι και να θυμηθούμε ότι πέρσι είχαμε τις, ε, βουλευτικές μας, τις κοινοβουλευτικές μας εκλογές και είχαμε το κίνημα που λεγόταν Vote for a Woman, ψήφισε γυναίκα. Και πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε ε, τις δημοτικές μας εκλογές με το ίδιο κίνημα, ψήφισε γυναίκα. Ήταν ε, πολλοί αυτοί που ήθελαν να ψηφίσουν μια γυναίκα, αλλά ψήφισαν πάντοτε την πρώτη του ψηφοδελτίου. Η πρώτη του ψηφοδελτίου θα εκλεγεί έτσι κι αλλιώ. Όταν λέμε ψήφισε γυναίκα, εννοούμε ψάξτε και λίγο. Ε, δηλαδή, άμα ξέρει κανεί τα ποσοστά που υπολογίζεται να πάρουν γυναίκε ε, με το εκλογικό αποτέλεσμα, καταλαβαίνει τι διαφορά μπορεί να κάνει ένα τέτοιο κίνημα. Ένα κίνημα που προβλήθηκε πολύ στο Facebook και το Twitter και εξελέγησαν περισσότερε γυναίκε στη Βουλή μα. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και για αυτό το παράδειγμα. Και ίσω θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε και βέλτιστη πρακτική για να το λαμβάνουν και άλλα κρατημέλη. Έχουμε μία ακόμη παρέμβαση από τη Γερμανία. Η κυρία Κχάνιχ. Ähm, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επανέλθω σε αυτά που είπε η κυρία Σουμάχερ για το πλέγμα αυτό των ε, δράσεων ε, τα προηγούμενα χρόνια. Πραγματικά είναι λυπηρό που το 2016 έπρεπε να γίνουν αυτές οι διαδηλώσεις των γυναικών, κυρίως στην Αμερική, ακριβώς επειδή η κατάσταση για τις γυναίκες στην, από την πολιτική σκηνή είναι πολύ δύσκολη. Εγώ ήμουνα σε μια διάσκεψη για το δικαίωμα των γυναικών και πολλά χρόνια συνεχόμενα βλέπαμε αυτές τις αποκλίνουσες εξελίξεις. Από τη μία είχαμε το θέμα της εκπαίδευσης για τις νέες γυναίκες στις αφρικανικές χώρες για παράδειγμα όπου βλέπαμε για χρόνια θετικές εξελίξεις και μέσω των εν μέσω πολέμων κτλ. Ε, βλέπαμε πόσα προβλήματα αντιμετώπιζαν τα κορίτσια κυρίως και βεβαίω ξέρουμε ότι από την άλλη η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την επιτυχία και οι γυναίκε πρέπει να μπορούν από μόνε του να καθορίζουν τη ζωή του. Όλα αυτά λοιπόν είναι άρρηκτα διασυνδεδεμένα μεταξύ του. Υπάρχει και η Σύνοδο ε, για το 2020, όπου πρέπει να συνδέσουμε τα θέματα αυτά, την διεθνοποίηση. Η, γυναίκα, η μέρα της γυναίκας δεν πρέπει να γιορτάζεται μία, μία μέρα το χρόνο μόνο. Εγώ είμαι μέλος όχι μόνο της Επιτροπής Γυναικών του Γερμανικού ε, Κοινοβουλίου, αλλά ξέρω ότι και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουν στο χέρι μας να διασυνδέσουμε ακόμη καλύτερα όλα αυτά τα δίκτυα, έτσι ώστε να έχουμε ένα μέλλον και στο ψηφιακό κόσμο για τις γυναίκες και στον πραγματικό κόσμο όμως. Και σε αυτό θα βοηθήσω όσο μπορώ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και να δώσουμε και πάλι το λόγο στην κυρία Σουμάχερ για να απαντήσει. Και μάλιστα μπορούμε να δούμε και τα αποτελέσματα των ερωτημάτων που θέσαμε. Μπορούμε παρακαλώ να τα δούμε στην οθόνη. Λοιπόν, ένα ερώτημα ήταν για το ποιες γυναίκες γνωρίζετε. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Η Αλίσσα Μιλάνου είναι πρώτη, αναφέρεται και στο δεύτερο ερώτημα. Είναι από τους ε, βασικούς ανθρώπους που ξεκίνησαν το κίνημα Me Μετά είχαμε την Μπάρμπαρα Νοβάτσκα, πολύ σημαντική φιγούρα για, την, ε, ε, για τις, για τις ε, διαδηλώσεις των, των μαύρων, για τις μαύρες γυναίκες, για τα δικαιώματα τα αναπαραγωγικά και τα δικαιώματα των γυναικών. Μετά έχουμε τρεις ακτιβίστριες από τα, από την, από τα κινήματα για, την, για τις ζωές των μαύρων γυναικών, η Σέρλ Σάντμπεργκ επίσης που αναφέρθηκε από την κυρία Σουμάχερ, με το Lean In, το hashtag, Έχουμε τη Rachel Sklar, επίσης τις απαντήσεις, που έκανε το ε, hashtag change the ratio και τέλος την, ε, επειδή βεβαίως οι περισσότεροι την ξέρατε, είναι η Μαλάλα, που δημιούργησε το hashtag we are silent και το σχετικό κίνημα. Πάρα πολύ σημαντική ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των κοριτσιών στην εκπαίδευση. Και το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με το πόσα άτομα απήντησαν εντός των πρώτων 48 ώρων μετά το πρώτο tweet της Αλίσσα Μιλάνο για το Me Too. Η πιο δημοφιλής ερώτηση είπατε ότι είναι το 1.200.000 άνθρωποι, αλλά η αλήθεια είναι ότι 5.700.000 άνθρωποι απήντησαν σε αυτό το tweet Οπότε βλέπουμε πραγματικά πόσο σημαντικό μέσο και πόσο ισχυρό μέσο είναι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να προωθηθούν τα δικαιώματα των γυναικών. Και η πιο δημοφιλής ερώτηση είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τα γυναικεία κινήματα των οποίων ηγούνται γυναίκες που χρησιμοποιούν την ε, πληροφορική. Ίσως η κυρία Σουμάχερ μπορεί να το ε, εντάξει στις ε, απαντήσεις της όταν θα απαντήσει και στα ερωτήματα από το πάνελ. Um, uh, Ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας για το ευρωπαϊκό μοντέλο, το πρότυπο το ελπίζω και εγώ να συμβεί και καλό θα ήταν όντω να δούμε ξανά τα θετικά στερεότυπα. Θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε γενικότερα τα στερεότυπα λόγω χάρη στα μέσα μαζική ενημέρωση, γιατί έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Εάν οι γυναίκε απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο από ότι. Ε, τώρα συμβαίνει και για τους άντρες. Το να βλέπουμε τους άντρες να σιδερώνουν, ας πούμε, θα κάνει μια διαφορά, ε, διότι ε, δουλεύουν ε, δυόμιση φορές παραπάνω οι γυναίκες ε, στις δουλειές ενός σπιτιού, στον οικοκυριό και για την κατάσταση των γυναικών θα είμαστε στη Νέα Υόρκη και στον ΟΗΕ τις ερχόμενες δύο εβδομάδες θέμα της Επιτροπής Γυναικών εκεί θα είναι οι γυναίκες στην Ήπεθρο. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν πλούσια και επικοδομητικά συμπεράσματα και η κυρία Κρόνιχ το ανέφερε, αλλά το ταξίδι μας συνεχίζεται. Θα πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη βασική ερώτηση, νομίζω, ναι, ότι το βασικό είναι να είμαστε δραστήριοι και δραστήριες. Να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνει το διαδίκτυο, αλλά και αυτές εκτός διαδικτύου, για να καλέσουμε κυβερνήσεις και άλλους φορείς να λογοδοτήσουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να εκφράσουμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας, τις επιθυμίες μας και από κοινού να εργαστούμε για μια καλύτερη κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ήταν ε, υπέροχο μήνυμα αυτό για να ολοκληρώσουμε και με αυτό το πάνελ και από τη δική μου την πλευρά πολλές ε, ευχαριστίες προς την Dagmar Schumacher από την UN ε, Women από το Νοιά και τις γυναίκες, είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια μπορούμε να κάνουμε βήματα πρόοδου και εκτό διαδικτύου και εντό, αλλά είδαμε και πολλέ επιθέσει και απειλέ κατά των γυναικών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη φαρέτρα μα, τα όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μα, και να αγωνιστούμε κατά αυτών των προσπαθειών. Να αγωνιστούμε για ισότερε κοινωνίε και κοινωνίε όπου όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Σα ευχαριστώ κυρία Σουμάχερ και θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Αντιπρόεδρο Παπαδημούλη, για τι καταληκτήριε παρατηρήσει του σε αυτή την ημερίδα. I ότι μπορώ να μιλήσω τη μητρική μου, τα ελληνικά, οπότε θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Παρακαλώ, βάλτε τα ακουστικά σας. Καλημέρα, σας λέγομαι Δημήτριος Παπαδημούλης, είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεταξύ των καθηκόντων μου είναι και τα θέματα της ισότητας και διαφορετικότητα ε, στο Ευρωκοινοβούλιο και νιώθω ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση διότι ε, πιστεύω ότι η διεκδίκηση των στόχων της ισότητας αφορά όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες που έχουν ε, ανοιχτό μυαλό και καταλαβαίνουν ότι είναι καλό για την κοινωνία να πετύχουμε τους στόχους της ισότητας και την κατάργηση των διακρίσεων. Σύμφωνα με μία μελέτη του OECD για να πετύχουμε τους στόχους της πλήρης ισότητας, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, χρειαζόμαστε 169 χρόνια. Είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσα πολλά χρόνια και για να το πετύχουμε αυτό γρηγορότερα χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Ε, κάποιος συνάδελφος είπε, ξέρουμε τις μελέτες, ξέρουμε τα στοιχεία, το θέμα είναι να κάνουμε περισσότερα. Στο Ευρωκοινοβούλιο το προσπαθούμε. Αν συγκρίνουμε την κατάσταση με το παρελθόν, έχουμε κάνει βήματα πρόοδου. Δεν μας αρέσει αυτή η μέθοδος γιατί οδηγεί σε μια επανάπαυση στο business as usual. Προτιμούμε να συγκρίνουμε τη σημερινή κατάσταση με τους στόχους που έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε την πλήρη ισότητα. Και συγκρίνοντας την σημερινή κατάσταση με το τι πρέπει να επιτευχθεί, το συμπέρασμα ότι χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά. Και η πολλή δουλειά, όπως προέκυψε και από τις συζητήσεις, δεν είναι μόνο δουλειά στην νομοθεσία ή στην εφαρμογή της νομοθεσίας, δεν είναι μόνο να φτιάχνουμε κανόνες, αλλά να επηρεάζουμε τα μυαλά και τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Να αντιμετωπίζουμε στερεότυπα. Για τους αριθμούς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 36% των μελών είναι γυναίκες, 36% των μελών επίσης του Προεδρείου είναι γυναίκες και 50% των μελών των Επιτροπών. Αλλά αν πάμε στους Προέδρους των πολιτικών ομάδων έχουμε μόνο μια γυναίκα και άλλη μια γυναίκα συμπρόεδρο σε ομάδα. Και αν πάμε στον Πρόεδρο και ο νυν Πρόεδρος είναι άνδρας και ο προηγούμενος Πρόεδρος είναι άνδρας. Άρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη συνεργασία και με τα εθνικά κοινοβούλια και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με τα Ινστιτούτα που μας βοηθούν πολύ, αλλά το πιο σημαντικό είναι το να ανοίξουμε ε, όσο το δυνατόν περισσότερο την επαφή μας με την κοινωνία. Στο διάστημα που έλειπα από εδώ, είχα πάει σε μια διπλανή αίθουσα για να συζητήσω με 300 περίπου νέα παιδιά που μετέχουν από το Στρασβούργο στο πρόγραμμα Euroscuola. Ε, τους μίλησα για την ημέρα της γυναίκας και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα ότι τα νέα κορίτσια που ήταν εκεί τα είδα πάρα πολύ μαχητικά στο να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει. Το πιο αισιόδοξο όμως στοιχείο ήταν ότι και τα γόρια που μίλησαν, τα νέα παιδιά, ήταν υποστηρικτικά αυτής της προσπάθειας θεωρώντας ότι είναι καλό για όλη την κοινωνία ε, να έχουμε μια κοινωνία με ίσα δικαιώματα και χωρίς διακρίσεις. Δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί και γι' αυτό ο στόχος της ισότητας και της διαφορετικότητας μπορεί να πάει χέρι-χέρι. Ε, αυτά θα ήθελα να πω γιατί έχουν ακουστεί πολλοί λόγοι για να μην μακρηγορήσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι να απολαύσετε και το διάλειμμα και το γεύμα που ακολουθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντιπρόεδρε Παπαδημουλή. Είμαι η Μέρη Χόνιμπολ, είμαι ε, μία από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής και έργο μου είναι να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ. Να σας ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχατε στα πάνελ και όλους τους ευρωβουλευτές και βουλευτές. Ήταν ε, μια εκπληκτική εκδήλωση και εμπειρία. Ευχαριστώ τους εθνικούς βουλευτές που έκαναν το κόπο και ήρθαν στις Βρυξέλλες. Ο δρόμος που μένει να διανύσουμε είναι μεγάλος, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μάθαμε σήμερα, να το προωθήσουμε και να συνεχίσουμε στο μακρύ μας αυτό έργο υπέρ της ισότητας, ότι κάποια στιγμή να είναι πράγματι οι άντρες και οι γυναίκες. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και γι' αυτό μας βοήθησε η σημερινή εκδήλωση. Ελπίζω αυτό να κρατήσετε από τη σημερινή μέρα. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξέρετε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι που ήρθατε. Ευχαριστώ τους οργανωτές της εκδήλωση και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για αυτή τη Διεθνή ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας.